Okay, Possiamo dare inizio, colleghi? Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζήτω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 13 της ημερησίας διατάξης. Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά. Κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ενιαίο κείμενο η συγκητή Σέρτζο Σιλβέστρης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο εισηγητή που θα παρουσιάσει την έκθεσή του για τον κανονισμό σε σχέση με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που επικεντρώνεται στα πιο αντιφατικά σημεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως θα ενημερωθήκατε όλοι, ζήτησα από τη γραμματεία μας να ετοιμάσει ένα τεχνικό σημείωμα τις περασμένες ημέρες ε, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς ε, σπόρων και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Πράγματι συχνά εσφαλμένα αναφέρεται κανείς ε, σε αυτή την αγορά ως αγορά στην οποία υπερισχύουν οι μεγάλες πολυεθνικές. Από το σημείωμα που εκπονήθηκε προκύπτει ότι οι περισσότερε επιχειρήσει ε, φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και σπόρων στι περισσότερε χώρε είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάλυση αυτού του φακέλου. Ο κ. Σιλβέστρη τώρα, στον οποίο θα δώσω το λόγο, θα το αναλύσει. συνέχεια μετά θα προχωρήσουμε στη συζήτηση με, το, με του συναδέλφου και μετά θα έχουμε και την ακρόαση με του εμπειρογνώμονε που έχουμε προσκαλέσει. Παρακαλώ, Σέλτζο Σιλβέστρη. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι, πριν να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας πούν τις απόψεις τους όσον αφορά τον τομέα σπόρων και φυτικών απορροφικού Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την έκθεση. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Έχει γίνει ανταλλαγή απόψεων στην ε, η Επιτροπή, αλλά μετά από την υποβολή του κειμένου είναι πρώτη φορά που ξεκινάμε συζήτηση. Φαντάζομαι και μάλιστα ελπίζω ότι πολλοί από εσά είχατε ήδη την ευκαιρία να εξετάσετε το σχέδιο έκθεση και τι τροπολογίε που υπέβαλα για την πρόταση τη επίτροπή και που θα σα παρουσιάσω σήμερα. Στο μεταξύ θα ήθελα να σα παρουσιάσω τα σημεία που θεωρώ κρίσιμα. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί καλή βάση εργασία. Ωστόσο, κάποιες έννοιες πρέπει να ευαθυνθούν και να συζητηθούν περισσότερο και ενδεχομένως να τροποποιηθούν εφόσον το θεωρήσει κατάλληλο αυτή εδώ η Επιτροπή. Τα σημαντικά σημεία είναι λίγα και σε αυτά επικεντρώνονται οι τροπολογίες μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλο το κείμενο το υλικό, εξειδικευμένο υλικό, niche material, ορίζεται από την Κομισιόν ε, ως ε, υλικό το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά από μικροεπιχειρήσεις, δηλαδή από μη επαγγελματίες, ε, οργανισμούς με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, με τζιρό κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αλλά αυτός ο ορισμός κατά την άποψή μου δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στον γεωργικό τομέα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχαν οι μόνιμες αντιπροσωπείες, τα στατιστικά στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το να εφαρμοστούν όλα αυτό που προτείνει η Κομισιόν, αυτός ο κανόνας δηλαδή που αφορά τον ίσματηριο, το ειδικευμένο υλικό που τίθεται σε κυκλοφορία στο εμπόριο από μικρές επιχειρήσεις με τζίρο κάτω των 2 εκατομμυρίων και με λιγότερο από 10 υπαλλήλου ε, αντιστοιχεί το 60% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και όλες αυτές θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Εξάλλου σας καλώ να λάβετε υπόψη σας τη μελέτη στην οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος Δεκάστρο η μελέτη που μας κατέφτασε χθε από τις εσωτερικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις διαστάσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα και στο μερίδιο αγοράς που κατέχουν. Εγώ για να βγούμε από αυτό το διέξοδο προτείνω να ε, ξαναορίσουμε εκ νέου το niche market, το ε, ειδικευμένη αγορά αναφερόμενοι όχι στην οντότητα των επιχειρήσεων παραγωγής αλλά στην οντότητα των παραγωγών που είναι περιορισμένες από άψη ποσοτική εκεί θα πρέπει να δώσει τον ορισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαδοχές ε, κατεξοδότηση πράξης ή θα πρέπει να ορίζονται βάσει τοπικών παραγωγών που μπορούν να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε στο εμπόριο ελεύθερα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν όσον αφορά αυτό το niche material, το ε, ειδικευμένο υλικό, μπορεί να επιληθεί με αυτόν τον τρόπο που μόλις περιέγραψα. Η δεύτερη πτυχή στην οποία θα ήθελα ε, επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας είναι το ετερογενές υλικό. Και αυτό δεν περιγράφεται λεπτόμερος από την Κομισιόν, παρότι είχε αρκετό χρόνο να ε, μελετήσει αυτόν τον ορισμό, ξεκινώντας από τις πρώτες Έρευνε μεταξύ εμπειρογνωμών ήδη από το 2007-2008. Ωστόσο, η Επιτροπή, παρότι χρειάστηκε 5 χρόνια για να εμβαθύνει αυτή την πτυχή, παρουσίασε ένα κείμενο το οποίο δεν συμμερίζονται ούτε καν οι ίδιοι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων οι οποίοι παραδοσιακά είναι εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να διευκολύνουμε αυτό τον ορισμό. Εγώ με την πρότασή μου προσπαθώ να παράσχω περισσότερη βεβαιότητα ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν ορισμό ο οποίο θα είναι πιο βέβαιο και θα το συμμερίζονται όλοι. Προσπαθώ δηλαδή να παρέχω περισσότερη βεβαιότητα στου παραγωγού του τομέα. Πρώτο ορισμό είναι τι εννοούμε με το αερογενέ υλικό Και εγώ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τους αδέλφους για κάποια μελλοντική ε, για κάποιο μελλοντικό συμβιβασμό για όσο λύσουν να συνεργαστούν έχω υποδείξει ότι το υλικό αυτό καταχωρείται με σύστημα παρόμοιο όπως αυτό που προβλέπεται ήδη για τις παλαιές ε, ποικιλίε. και αυτό είναι ένα σύστημα προϋποθέσεις πολύ πιο ελαφρές ε, από, την αρχική, από το, αυτές του αρχηγορισμού κοστίζει λιγότερο και βασίζεται σε γνώσεις που αποκτήθηκαν με πρακτική εμπειρία κατά την καλλιέργεια, την αναπαραγωγή και τη χρήση. Εγώ έχω την εντύπωση, έχοντας συζητήσει με τους εμπειρογνώμονες ε, του τομέα, ότι θα υπάρξει δυνατότητα να επιτευχθεί συνένεση με όλους τους συναδέλφους. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που συγκεντρώνει και τις περισσότερες τροπολογίες στο σχέδιο εκθεσής μου σχετίζεται με την αξία, με την VCU, την αξία καλλιέργειας και χρήσης. Αυτή η έννοια που αποτέλεσε αντικείμενο της παράθεσης πολλές φορές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξεταστεί. Όπως εξήγησα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας, η Κομισιόν στην πρότασή της δημιουργεί μια διάκριση μεταξύ ικανοποιητικής αξίας για καλλιέργεια, η χρήση, και της βιώσιμης αξίας για την καλλιέργεια. Στην τρέχουσα νομοθεσία δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ ικανοποιητικής και αηφόρου αξίας. Γι' αυτό το λόγο στην εκθεσή μου προτείνω να συνενώσουμε του δύο σε μία, σε μία αυτή η αξία βάσει τη οποία αξιολογείται η εγκυρότητα μια νέα ποικιλία, έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, όπω μαρτυρείται από διάφορε συναντήσει που είχα εγώ με διάφορου ενδιαφερόμενου και εμπειρογνωμόνε στο τομέα. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγο να τροποποιήσουμε σήμερα αυτό το καθεστώ, το οποίο κατά την άποψή μου θα οδηγούσε σε στόχο αντίθετο από το στόχο τη προτάση αυτή. Αυτή η πρόταση, Αυτό ο νέο κανονισμό, έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους. Ε, και μια τέτοια πρόταση θα διπλασίαζε και μέσω μιας διάκριση που δεν είναι περιττή. Υπάρχει κίνδυνο να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία και τι δαπάνε. Για αυτό το ζήτημα λοιπόν ήθελα να προσθέσω ότι η Κομισιόν στο αρχικό κείμενο προβλέπει ότι το VCU θα πρέπει το ικανοποιητικό VCU πρέπει να μετράται σε κρατικό επίπεδο και το, το βιώσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον ένα ενιαίο VCU ε, θα είμαστε στο επίπεδο των κρατών μέλων που ούτως ή άλλως θα πρέπει να εξετάσουν τις πτυχές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα πρέπει να εποπτεύει ώστε να, να βεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται όλοι με τα πρότυπα ποιότητα. Μετά από μια πρόσφατη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ότι για το ζήτημα αυτό έχουμε συμφωνήσει. Και όσον αφορά το ενίο VCU, την ενιαία VCU, και η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνενέσει σε σχέση με τα όσα προτείναμε. Ένα άλλο θέμα είναι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς, για καλοπιστικούς σκοπούς. Στην τρέχουσα διατύπωση του κειμένου, ορισμένα ήδη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για καλοπιστικούς σκοπούς, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διατροφικούς σκοπούς, όπως ε, ε, ο το, θα πρέπει λοιπόν να γίνεται στον κανονισμό μια διάκριση χρήσεων. Σκοπός μου λοιπόν είναι να ζητήσω λιγότερο αυστηρούς κανόνες και επίσης πρέπει να δούμε και την αντιστοιχία με τις τρίτες χώρες ε, και ευχαριστώ την Κομισιόν ε, έχουμε ζητήσει πολλές φορές να εξεταστεί τη ισοτιμία ε, των προτύπων για τα εισαγόμενα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η τρίτη χώρα με την οποία, από την οποία εισόγουμε δεν έχει τους κατάλληλους κανόνες, θέλουμε στο πλαίσιο συμφωνιών για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ε, να υπάρχει μια συμφωνία για τα πρότυπα αυτά ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι 12 οδηγίες ε, της Ευρώπης, ε, οδηγίες δεν καλύπτουν εξαγωγή του υλικού όλο το πακέτο για ε, την υγεία και την ε, προστασία των φυτών και των ζώων ε, είναι τέτοιο που προτείνω να ενημερώσουμε όλη αυτή την νομοθεσία. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις ισοτιμίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών που παράγεται σε τρίτες χώρες, πιστεύω ότι οι εκτελεστικές πράξεις που ζητάει η Κομισιόν πρέπει να γίνουν τις πράξεις, ώστε να μπορεί να δώσει την άποψη της σε, για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό για το κοινοβούλιο. Για να αφήσω χώρο τώρα για συζήτηση και για τις παρεμβάσεις των εμπειρογνώμων που θα ακούσουμε όλοι με μεγάλη προσοχή. Κάποια τελικά σχόλια θα ήθελα να κάνω για τις εξουσίες που εκχωρούνται στην Κομισιόν. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το παράδειγμα 1 του κειμένου που ορίζει τον κατάλογο των ειδών που θα εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού ζήτησα εγώ αυτό το παράδειγμα 1 και το 9 για τα δασικά πολυπρεσιαστικά υλικά να τροποποιηθούν να τροποποιούνται μέσω ε, τακτικών νομοθεσιών και όχι μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ λοιπόν και τη συναδελφογή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος που συμμετείχε και στη συνάντηση σκιωδών γιατί πιστεύω ότι το κείμενο της ήταν πολύ σημαντικό το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Για να κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι, να επαναλάβω ότι είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, να συζητήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε ώστε να ορίσουμε τι οδό θα ακολουθήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της, τους συμβούλους, τους κοιόδης, τους βοηθούς τους και το προσωπικό του γραφείου μου για την υποστήριξη τους σε αυτό το έργο το οποίο ξεκινάει πλέον επίσημα. Πιστεύω ότι με τη σύσταση προτάσεων και όχι ιδεολογιών ε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε συνεργαζόμενοι με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό. Ευχαριστώ όλους. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε τον κύριο Σιλβέστρη. Σας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν πολλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε τον Μάρτιν Όσλινγκ και μετά Κάδεμβαχ. Μάρτιν. <clears throat> ναι, θα έλεγα ευχαριστώ τον κύριο Σιλβέστρη για την προθυμία περαιτέρω τροπολογίες να εξεταστούν, διότι θα είναι αναγκαίο πιστεύω να γίνει αυτό. Το σχέδιο όπως το έχουμε μπροστά μα δεν μπορεί έτσι να ολοκληρώνει το θέμα. Έχουμε και κάποιες επικρίσεις, κάποια σημεία που πρέπει κάποια πράγματα να πούμε. Αυτά που την τελευταία φορά συζητήσαμε σχηδός Για παράδειγμα το δικαίωμα των γεωργών, το προτέρημα των γεωργών. Μας ρώτησαν συγκεκριμένα στο σχέδιο κανονισμού δεν θα μπορούσε να ρυθμιστεί καλύτερα ότι τώρα δεν πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με το, τους γεωργούς με ένα νομικό κείμενο, να αφήσουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας και ελαστικότητας δεν έγινε αυτό. Δεν συμπεριλήφθηκε αυτό το οποίο αφορά την βιολογική γεωργία και τα κριτήρια σχετικά. Τα κριτήρια για τον, τους βιολογικούς σπόρους δυσχεραίνουν τα πράγματα σύμφωνα με, α, άλλες, με άλλα είδη τα οποία έχουν διευκολύνσεις, ενώ εδώ δυσχεραίνονται τα πράγματα, δεν δίνονται απαντήσεις, αντίθετα διαγράφονται εξαλείφονται δυνατότητες ε, να εκμεταλλευτεί κανείς κάποιες μικρές αγορές, ε, νης. Δεν είμαι υπέρμαχος του να υπάρχουν τέτοιου, τέτοιου είδους ε, αποκλειστικότητες για προϊόντα ή αγορές. Αλλά όμως περιορίζουμε περαιτέρω το πλαίσιο εφαρμογής. Δεν ξέρω γιατί. Φοβούμαι ότι στο τέλος θα οδηγούμαστε σε περισσότερες ρυθμίσεις και διατάξεις και μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και στο τέλος τέλος όσον αφορά το προκυπευτικά και τα βότανα με έναν τέτοιο κανονισμό είναι τα πράγματα πολύ δυσνόητα. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει πια κανείς τι θα γινόταν σε σχέση με τους σπόρους. Τέτοιου είδους ε, τομείς να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο ελέγχου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει κάτι τέτοιο και ακόμα και για τις ε, μεγαλύτερες ας το πούμε φυτικές ασθένειες δεν απειλούν αυτές, αυτά τα είδη. Ίσως κάτι άλλο, σε κάτι άλλο οφείλεται αυτή η κατάσταση. Ίσως μπορείτε να το απαντήσετε. Είπατε μετά θα υπάρξει εξαίρεση για περιφερειακά είδη και ποικιλίε. Εντάξει, περιφερειακές ποικιλίε. Είναι δύσκολα τα πράγματα να καθοριστούν αυτές οι περιφερειακές ποικιλίε από πλευράς τοπίου και περιφέρειας ε, περιοχής και περιφέρειας ε, θα διαφοροποιούνται αυτά ή πώς. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ερμηνείας εδώ. Θα πρέπει να βελτιωθούν πολύ τα πράγματα με κάθε σαφήνεια. Αν θέλουμε να είναι εξαιρέσει κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν κατανοώ όμως είναι το ότι κατά τα άλλα δεν θα έχουμε ετικετοποίηση και διαφοροποίηση και αυτό για την βιολογική γεωργία έχει συγκεκριμένη σπουδαιότητα και για τις διάφορες τεχνικές παραγωγής σπόρων, CMS. Δεν είναι κάτι που δεν είναι αμφίσιμο, που δεν έχει, ας το πω έτσι, δεν ασκούνται επικρίσεις. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Υπάρχουν πολλά σημεία που σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής βρισκόμαστε πιο πίσω από το απαιτούμενο επίπεδο. Έλπιζα ότι ο εισηγητής θα μπορούσε να διευκολύνει τα πράγματα, να τα διευκολύνει για τους γεωργούς και κάποιους τομείς να τους εξαιρέσει τελείως από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Διότι ήδη την πρώτη φορά άσκησα επικρίσεις. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποια μεγέθη και στοιχεία ότι υπάρχει λέει τεράστια βιοπικιλότητα σε σχέση με τους σπόρους. Έχουμε ναι, με μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με αυτά. Σωστό. Αν δει κανεί όμως ε, το ευρύτερο πλαίσιο τότε εκπλήσεται και κάποιες επιχειρήσεις που έχουν όνομα στην αγορά αλλά δεν είναι πλέον αυθύπακτες αυτοτελείς. Δεν μπορούν εκείνες να καθορίσουν τις εξαιρέσεις σε σχέση με τους σπόρους. Και η συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί και στην Ευρώπη στρεβλώνεται. Θα έχουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη που αυτή η αγορά πλήρως θα τεθεί υπό έλεγχο κάποιον. Κάπως πρέπει να αντισταθούμε, να μην γίνει κάτι τέτοιο και σε σχέση με τις απαντήσεις σε αυτά τα θέματα από τον εισηγητή πρέπει να δοθούν απαντήσεις, βιοπικιλότητα, εξαιρέσεις και εδώ αντί να προχωρήσουμε έτσι έχουμε περιορισμούς και ένα δίσκαμπτο πλαίσιο. Δεν είναι αυτή η ενδεδειγμένη απάντηση. Είμαστε όμως πρόθυμοι να ξαναπεράσουμε στην εξέταση αυτών των θεμάτων ελπίζοντας ότι κάποια πράγματα μπορούν να συμπεριληφθούν και να βελτιώσουν τις προτάσεις. Τα βλέπουμε ίσως με πιο κριτικό μάτι σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπής από άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν, Κάιν, Κανεμπάκ και μετά Ρόντους. Σας ευχαριστώ θερμά Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτόν τον κανονισμό για την παραγωγή αναπαραγωγικού φυτικού υλικού και την διάθεση στην αγορά για παράδειγμα σε σχέση με τους σπόρους στην Ευρώπη ξεκίνησε με βάση αυτή την πρόταση ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων. Είμαι υπέρ αυτή η συζήτηση σήμερα να συνεχιστεί βέβαια, διότι τα σπόροι και το αναπαραγωγικό υλικό είναι τα θεμέλια των τροφίμων μας. Όμως από την άλλη πλευρά να ανησυχώ γιατί σε μια εβδομάδα, 4 Δεκεμβρίου, θα εκπνεύσει η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για ένα τόσο περίπλοκο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που έχει και τόσο ε, σύνθετο χαρακτήρα θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο. Με το ρόλο μου ως κοιόδους εισηγήτριας ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα της έκθεσης του κυρίου Σιλβέστης. Μια ολόκληρη σειρά συζητήσεων έκανα και εργαστήρια, workshops έγιναν στα οποία συμμετείχα. Και αν δούμε τώρα τα επιμέρους σημεία που σε σχέση με την βελτίωση για το status quo δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ μια τέτοια βελτίωση. Το αντίθετο, βλέπω μια επιβάρυνση γραφειοκρατική, μια γραφειοκρατική θα έλεγα ε, περιπλοκή που δυσχεραίνει τα πράγματα. Θα έπρεπε να μην γίνει αυτό. Η ε, σύγκριση διάφορων οδηγιών σε ένα κανονισμό μπορεί να θεωρείται ή να αποκαλείται απλούστευση. Όμως για το πεδίο εφαρμογής της, ε, ε, του πλαισίου αυτού από 250 είδη να επεκταθούμε σε όλα τα είδη από πλευράς ποικιλότητα δεν είναι απογραφειοκρατικοποίηση και τι θα γίνει με την απλούστευση αυτή. Μεγαλύτερη επιβάρυνση γραφειοκρατική από πλευρά των κρατών μελών. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Και το τι γίνεται σε σχέση με ε, τις ε, ζωοτροφές. Ε, το πακέτο αυτό βρίσκεται υπό τον τίτλο «Εφιέστεροι κανόνες για ασφαλέστερα, ασφαλέστερα τρόφιμα». Πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε τα πράγματα λοιπόν. Εμείς ως Ευρωβουλευτές ελπίζω ότι μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή τη στάση σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής ε, αυτού του κανονισμού σε σχέση με τις προηγούμενες οδηγίες. Διότι εδώ υπάρχει επικάλυψη. Τα κράτη-μέλη θα απολέσουν τους αναγκαίους ε, χώρους και περιθώρια που είναι αναγκαία για αυτά, για το πεδίο εφαρμογής. Θα είμαστε πολύ πιο δίσκαμπτοι. Ο κανονισμός πρέπει να περιορίζεται στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό για τρόφιμα και ζωοτροφές που ε, οδηγούνται στην εμπορία. Πρόκειται για μια ρύθμιση της αγοράς. Δεν μπορεί εμπορικές δραστηριότητες να τις επικαλύπτει. Δεν είναι αυτό το νόημα αυτού του κανονισμού. Δυστυχώς αυτός ο κανονισμός στους επαγγελματίες πρέπει να περιορίζεται. Σε σχέση με αυτούς δηλαδή που εμπορεύονται επαγγελματικά αυτούς τους σπόρους. Για όλους τους άλλους θα πρέπει όλοι οι άλλοι να εξαιρεθούν, οι οποίοι δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα αυτή τη δραστηριότητα. Δεν έχει νόημα να απαιτεί ρυθμίσεις και διατάξεις αυτός ο κανονισμός για 300.000 είδη και να επιβαρύνονται τα πράγματα. Ενώ έχουμε 250 είδη τα οποία καλύπτονται από τις οδηγίες σήμερα. Ανεπαρκής είναι και η όρη για την βιοπικιλότητα και για το γενετικό υλικό, φυτικό γενετικό υλικό. Και από πλευράς προλαλήσαντος αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε εδώ να αντισταθούμε στην επιβάρυνση τη γραφειοκρατική. Συγκεκριμένες προτάσεις, η απλουστευμένη αδειοδότηση, η επίσημη δηλαδή ε, αναγνώριση για καταχώρηση και αδειοδότηση, ο κάθε ένας που οδηγείται σε γεωγραφικούς περιορισμούς ή ιστορικούς περιορισμούς πρέπει να παραδεχτεί ότι πρέπει να καταργηθούν τέτοιου είδους περιορισμοί. Είναι αντιπαραγωγικό να έχουμε ένα τέτοιο στενό πλαίσιο και για τους ε, σπόρους ε, ε, των φυτών και για τον περιορισμό σε σχέση με ειδικέ ποικιλίε θα έπρεπε χωρίς περιορισμούς και με δίκαιο πλαίσιο να μπορούν να διοχετεύονται στην αγορά. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει την συμπίκνωση, την επικέντρωση σε λίγα χέρια της αγοράς. Βλέπω ότι δεν είναι η βιοπικιλότητα η οποία διασφαλίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν δούμε τη γαλλική αγορά, διαρωτάται κανείς Πώς γίνεται κάποιες λίγες εταιρείες να έχουν το λέγει, να έχουν το πάνω χέρι και να έχουν δεσπόζοντα ρόλο στην αγορά. Μια άλλη εικόνα λοιπόν αναφύεται αν τα δει κανεί έτσι. Στόχο μα πρέπει να είναι το δυνατόν περισσότεροι εμπλεκόμενοι ω παίκτε να συμμετέχουν στην αγορά. Αναφέρθηκε ότι κάποιοι λίγοι έχουν τεράστια επιρροή σε 70% της αγοράς. Και για τους καταναλωτές το ευρωβαρόμερο το, το δείχνει. Θέλουν ποικιλομορφία οι καταναλωτές, όχι μόνο για λόγους βιοποικιλότητας αλλά επειδή για λόγους γεύσης, επειδή προτιμούν κάποιες γεύσεις, θέλουν να υπάρξει αυτή η διασφάλιση. Έχουμε πάρα πολλά είδη πατάτας για παράδειγμα, που διοχετεύονται στην αγορά και σε λίγες μέρες ε, εξαντλούνται τα ε, φύτα αυτά, τα προϊόντα αυτά. Δηλαδή ο κόσμος τα αγοράζει αμέσως. Πρέπει να δούμε πώς τα απορροκυπευτικά αυτού του είδου τα προϊόντα θα διοχετεύονται με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά. Οι καταναλωτέ πρέπει να αποφασίζουν τι θα καταναλώνουν, αν θέλουν κάποια περιφερειακή ποικιλότητα που προτιμούν και θέλουν να αγοράσουν. Έτσι λοιπόν μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών θα κατατεθούν για να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα. Και έτσι αυτή τη σκέψη βιοποικιλότητας θα μπορούσαμε να την διασφαλίσουμε, να την κατοχυρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κάρεν και μετά ο σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω τώρα εδώ να κάνω κάποιες δηλώσεις και να μακρηγορήσω. Πέντε ερωτήματα έχω που θα ήθελα να διατυπώσω. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Σιλβέστρης για το έργο που επετέλεσε και την έκθεση που μας παρουσίασε. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Σε σχέση με κάποια προϊόντα ή νίσο όπως αναφέρεται. Δεν το κατανόησα απόλυτα. Μπορείτε ίσως να το απαντήσετε. Είναι δυνατόν, λέει η ερώτηση, παλαιά προϊόντα και είδη με βάση μια τέτοια διαφοροποίηση με την, ε, τον προσδιορισμό, επίσημο προσδιορισμό να διοικητεύονται στην αγορά. Ένα δεύτερο ερώτημα. Διασφαλίζεται ότι η αδειοδότηση ειδών και ο έλεγχος της ποιότητας των σπόρων σε κρατικά χέρια θα παραμείνουν. Αυτή η έλεγχη. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Για τους συναδέλφους ε, τα κριτήρια για την, ε, τους ελέγχους ε, που αναφέρθηκαν. Ερώτηση σε σχέση με αυτό. Ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με την μείωση και την, ας το των ε, επιβαρύνσεων των παραγωγών. Φυσικά με την εγγύηση ότι αυτοί οι σπόροι θα διασφαλίζονται στην ποιότητά τους ε, για όλους ε, σε υψηλά επίπεδα. Σημαντικό είναι για μένα και το θέμα των γενετικά τροποποιημένων ειδών. Υπάρχει δυνατότητα ίσως και τα ηχέγγυα ώστε να έχουμε ελεύθερες από γενετικές τροποποιήσεις τέτοιους σπόρους. Πώς θέλετε να το διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί αυτό. Τελευταία ερώτηση. Είναι δυνατόν ήδη που η προστασία τους έχει λήξει να συνεχίσουν να υφίστανται, να είναι διαθέσιμα στην αγορά. Να εγγυηθούμε δηλαδή ότι θα είναι δυνατόν τα παλαιότερα ήδη, οι ποικιλίε να μπορούν να βρίσκονται στην αγορά. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις θα ήταν πολύ καλό. Δεν θα έπρεπε να θέσω κάποιες τροπολογίες. Αλλιώς θα σας επιβαρύνω με τροπολογίες που θα καταθέσω αν δεν απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και Έχουμε τον Άγνιο τώρα και μετά τον Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω λάβει πολλά γράμματα πάνω στην οδηγία αυτή τη λεγόμενη οδηγία για τους ε, σπόρους, για τα κυπευτικά και η Κομισιόν δεν θα μπορούσε να έχει κάνει μεγαλύτερο αυτογκόλ πριν, έξι μήνες πριν τις ε, ευρωεκλογές. Πολλοί κόσμος στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τώρα δεν ανησυχούσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα βλέπουν να επηρεάζεται η ζωή τους. Και ξέρετε ότι λέμε ότι το σπίτι του Άγγλου είναι ε, το παλάτι του και αυτό περιλαμβάνει και τον ε, κήπο με τα οποροκυπευτικά και ε, ειλικρινά σας λέω δεν τους αρέσει καθόλου η οδηγία αυτή και μπορεί να αναρωτιέστε ποιο είναι το σκάνδαλο που οδήγησε σε αυτήν την νομοθεσία. Είδαμε κάποια νέα νόσο των φυτών που προέκυψε από τον κήπο κάποιου, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Ε, πούλησε κανείς σε κάποια λαϊκή αγορά κάποια ντομάτα ή κάτι τέτοιο που να οδηγήσει σε μεγάλη ε, σε κάποια εξάπλωση μιας ασθένειας ε, στην χώρα. Από ό,τι γνωρίζω όχι. Έχει να κάνει με την επιθυμία της Κομισιόν να νομοθετεί πάνω σε κάθε τομέα της ζωής μας και υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι μεγάλος αριθμός σπόρων και αναπαραγωγικού υλικού μπορεί να εξαφανιστούν από την αγορά και έχουμε εδώ ένα προηγούμενο πριν ένα-δύο χρόνια ή μπορεί πιο ε, παλιά. Ε, μετά την εκλογή μου πάντως είχαμε νομοθεσία σχετικά ε, με τα φυτοφάρμακα και κάποιοι παραγωγοί αποφάσισαν να σταματήσουν να παράγουν τα φυτοφάρμακα αυτά λόγω του κόστους καταχώρησής του. Ένα από τα φάρμακα αυτά καταργήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα να δούμε τις στέρες να εξαπλώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, στην ε, εξοχή της ε, Αγγλίας. Και πιστεύω ότι η παρούσα νομοθεσία θα οδηγήσει τις εταιρείε ώστε να μην βρίσκει ο κόσμος τους πόρους που θέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντόρφμαν και μετά Πέτριαρ. Herbert. Κύριος Ντόρφμαν, ευχαριστώ. Ιταλικά θα μιλήσω Ιταλικά. Έχοντα, ακούσει τόσο είπε ο συγγετής μας, ο Σιλβέστρο και οι επόμενοι συνάδελφοι, όσον αφορά τους ορισμούς, ε, δεν έχουμε διαφορετική γνώμη ιδιαίτερα. Όλοι συμφωνούμε ότι όσοι καλλιεργούν ή παράγουν σπόρους ή φυτά ή αναπαραγωγικό υλικό όχι επαγγελματικά εξαιρείται από αυτή την οδηγία. Αλλά εγώ, δια, αυτό τον κανονισμό, συγγνώμη, αλλά διαβάζοντα το άρθρο 2 μαζί με το άρθρο 3, μου φαίνεται ότι αυτή είναι η πρόταση, επειδή το άρθρο 2 λέει ότι ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για μη επαγγελματίες ε, στον τομέα της αναπορρογής των φυτών. Ένας λοιπόν απλός γεωργός που ανταλλάσσει σπόρους με τον γειτονά του ή μια ομάδα ανθρώπων που το κάνει ως χόμπι εξαιρείται. Αυτό θα πρέπει να οριστεί καλύτερα ώστε να καταλάβουμε καλά τι εννοούμε. Ωστόσο εγώ έχω την εντύπωση ότι όλοι συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι δεν θέλουμε να μην πλήξει ο κανονισμός αυτός ε, όποιον δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα αυτόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μου φαίνεται ότι είναι εξειδικευμένε αγορέ. Τα εξειδικευμένα είδη. Γιατί εγώ συμφωνώ με τον συναδελφό κύριο Σιλβέστρη, διότι η εξειδικευμένη αγορά έτσι όπω ορίζεται από την Κομισιόν δεν μπορεί να είναι εξειδικευμένη, διότι το γεγονό ότι μια επιχείρηση είναι μικρή δεν σημαίνει ότι δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένη αγορά. Για παράδειγμα, ε, ε, εγώ έρχομαι από μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλές μιλιές, παράγουν πολλά μιλά το χρόνο. Ο κάθε φορέας παραγωγής έχει λιγότερο από 10 υπαλλήλους και λιγότερο από 2 εκατομμύρια τζίρο. Ωστόσο όλοι παράγουν φυτά που πρέπει να πιστοποιηθούν αναγκαστικά διότι όποιος αγοράζει ένα μήλο, αγοράζει μια συγκεκριμένη ποικιλία, πρέπει να είναι σίγουρος ότι αυτό είναι το φυτό. Δεν μπορεί να ρισκάρει να αγοράσει ένα οποιοδήποτε φυτό μη αναγνωρίσιμο, μη επιστοποιημένο, το οποίο μετά από τρία ε, χρόνια θα, παράσει διαφορετικό προϊόν από αυτό που είχε υποσχεθεί. Η εξειδικευμένη αγορά λοιπόν δεν μπορεί να βασίζεται στο μέγεθος ε, Ενό αγροκτήματο, διότι ακόμα και αν έχει λιγότερου από 10 υπαλλήλου και κάτω των 2 εκατομμυρίων ε, τζίρο μπορεί να, έχει, να παράγει μια κλασική ε, ποικιλία μήλων. Δεν εξαρτάται λοιπόν από το μέγεθος ε, του αγροκτήματο. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με τον Σιλβέστρη ότι πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο ορισμό. και ίσως και η συζήτηση που θα ακολουθήσει να μπορέσει να μας βοηθήσει. Θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι εξειδικευμένη αγορά που για μένα θα πρέπει να εξαιρείται από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ωστόσο εγώ είμαι πεπισμένος επίσης ότι, ότι το σημαντικότερο που πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι Ποιο αγοράζει το σπόρο, οποιοδήποτε ε, γεωργό αγοράζει το σπόρο, ε, πρέπει να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι αγοράζει. Έχει δικαίωμα να αποκτήσει την ποικιλία την οποία ήθελε να αγοράσει. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον το υλικό που έχει αγοράσει είναι πιστοποιημένο. Ε, έτσι, θα, αυτή η ποικιλία εξειδικευμένων αγώνων θα πρέπει να αποτελέσει το δικαιώμα διαφορετική διαχείριση. Πέτερ Γιάρ τώρα και Τζορτζ Λάιον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή που με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αφορά, ασχολείται με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα, ζήτημα και αυτό αφορά και τα μηνύματα τα οποία μας απεστάλησαν. Και θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα σε σχέση με την αποστολή μηνυμάτων και τα όσα μας είπαν οι καταναλωτές. Το πρώτο συνεχίζει αυτά που αναφέρθηκαν πιο πριν. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε εκείνους που εφαρμόζουν οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι δηλαδή ας το πω έτσι σε αυτή τη δραστηριότητα και θέλουν τη διατήρηση αυτού του ομογενοποιημένου υλικού. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει φυτικούς σπόρους πρέπει να ξέρει ποιοι είναι, τι είδου είναι αυτοί και να είναι ομοιογενές προϊόν και όχι ετερογενές προϊόν. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις που να διασφαλίζεται η ποιότητα. Η φυτική σποροπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικά θα έχανε σε ποιότητα αν δεν λαμβάναμε αυτό υπόψη. Δεύτερον, η διατήρηση παλαιότερων ποικιλιών με νήσε τις αγορές ε, συγκεκριμένου πεδίου, περιφερειακές αγορές ε, και πεδία εφαρμογής εξειδικευμένα. Πρέπει να δούμε τον ορισμό. Τι είναι περιφερειακή αγορά. Κάποιοι χαρακτηρίζουν την Ευρώπη περιφερειακή αγορά. Και πάνε τα πράγματα πολύ γρήγορα έτσι, όταν τα απλουστεύουν έτσι. Και όταν έχουμε κάποιο παλαιό, κάποια παλαιά ποικιλία και υπάρχει επιτυχία, τότε κάποιο επιχειρηματία δεν θα αντισταθεί όπω θα έπρεπε στον πειρασμό να υπεκτείνει και να διευρύνει διαρκώ ε, το πεδίο εφαρμογής αυτής της περιφέρειάς του και θα το επεξέτεινε διαρκώς. Και εγώ είμαι υπέρ της διατήρησης των παλαιών ποικιλιών. Και χαίρομαι και θα χαιρόμουν αν μπορούν αυτές να καλλιεργούνται στο μέλλον. Αλλά εδώ δεν πρέπει να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Να έχουμε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Ένα διαφορετικό πύχη με διαφορετικά μέτρα και σταθμά να μετράμε και να σταθμίζουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην υπάρξει κάποια παράλληλη τροχιά που θα ανοίξει να κινηθούμε παρεκκλίνοντας από αυτούς τους στόχους. Και για τους οικολογικούς ε, γεωργούς θα πρέπει ομοιογενές υλικό να είναι αυτό για τους σπόρους ε, που καλλιεργούν. Δεν κατανοώ την ε, ένταση στη συζήτηση. Λένε ότι η οικολογική γεωργία, οι γεωργοί που ακολουθούν οικολογικές αρχές παίρνουν στα χέρια τους τέτοιες πρωτοβουλίες με ομοιογενεί τέτοιες, τέτοιες ποικιλίε. Επανερχόμαστε στο παλαιό πρόβλημα τι είναι ακριβώς περιφερειακή αγορά και τι είναι πεδίο, εξειδικευμένο πεδίο εμπορίας ε, ή εξειδίκευσης. Και μπορώ σε σχέση με τα μηνύματα που μας ε, στάλησαν να πω το πιο συχνό είναι πώς μπορούμε να τραβήξουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ επαγγέλματος ε, και χόμπι. Δηλαδή βλέποντας για παράδειγμα, δίνοντας για παράδειγμα κάποιος στο γείτονα σπόρους, ε, δεν θα είναι επαγγελματία. Έτσι, αυτή η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να είναι σαφή για να ισχύει για όλου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι σαφέστερο λοιπόν αυτό το διαχωριστικό, αυτή η διαφοροποίηση από ότι στην πρόταση της Επιτροπή. Το επόμενο, αγαπητέ εισηγητά, με την σημερινή πρόταση τι γίνεται. Δυστυχώ έχουμε και μια διαφορά σε σχέση με τα διάφορα φυτά λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη τις διαφορές. Κάποιοι έχουν δασοκομικές, δασοπονικές δραστηριότητες, τα δάση πρέπει ξεχωριστά να αντιμετωπίζονται ε, και διαφορετικά έχουμε οποροκυπευτικά, δημητριακά, θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση και όχι να συγχέονται όλα γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πέτερ, George Lyon και μετά Στάντλερ. George. Uh, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Σιλβέστρηση για την έκθεσή του. Νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σε διάφορους τομείς. Και ελπίζω ότι οι ενδεχόμενες τροπολογίες θα βασιστούν πάνω στη δουλειά που έχει ήδη κάνει. Άλλωστε, αφατηρία για όλα αυτά είναι ότι το σύστημα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να ε, μπορεί να βοηθήσει στο να θρέψουμε την Ευρώπη και να μπορέσουμε να εξάγουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους ε, καταναλωτές, ε, τους ε, γεωργούς, τους καλλιεργητές. θέλουμε λοιπόν ό,τι αναφέρεται στο, στη συσκευασία να είναι αλήθεια, να μην υπάρχουν οι ισχυρισμοί. ψευδείς, διότι στο κάτω-κάτω Ο Γεωργός ε, πρέπει να ξέρει τι μπορεί να προσδοκεί όταν ε, αγοράζει κάποιους ε, σπόρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά του. Και ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία στους μικρούς εξειδικευμένους καλλιεργητές, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι παρεκκλήσεις αυτές, ε, οι προσαρμογές ε, να μην επιτρέψουν στις εταιρείε ε, να παρακάμψουμε την υποχρέωση περί καταχώρησης. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Η ουσία της συζήτηση λοιπόν είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό και πώς θα ορίσουμε αυτούς τους εξειδικευμένους καλλιεργητές. Και είμαι βέβαιος ότι τίθεται και όλο το θέμα του ποιος πληρώνει τα δικαιώματα. Όπως είπε ο συνάδελφός μου ο κύριος Ντόρφμαν ε, πριν λίγο, το ε, να ορίζεται αυτό το εξειδικευμένο πεδίο μέσω του αριθμού των ε, υπαλλήλων και του μεγέθους της εταιρείας δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλός τρόπος. Βρίσκω πολύ περίεργη γενικά αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες ώστε να την ε, τροποποιήσουμε, όπως άλλωστε ήδη έχει κάνει ο κύριος Σιλβέστρης. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε μόνο κάποιους λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μικρότερων ε, επιχειρήσεων ε, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και σε αυτές να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν ε, στην αγορά. Η ιδέα ότι στην αγορά δεσπόζουν οι τρεις-τέσσερις μεγάλες εταιρείες είναι λανθασμένη. Επίσης θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η βιοπικιλότητα είναι κάτι που ζητούν οι καταναλωτές. Ε, ε, ε, ότι η βιοπικιλότητα εξαρτάται από τους καταναλωτές ε, και όχι από τους γεωργούς. Ε, οι γεωργοί καλλιεργούν αυτά που ζητάει η αγορά. Η βιοπικιλότητα λοιπόν εξαρτάται από την ζήτηση των, από πλευρά των καταναλωτών. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα στην αγορά. Κανένας γεωργός δεν θα καλλιεργήσει κάποια ποικιλία επειδή έτσι του αρέσει. Αν αρχίσει να καλλιεργεί περίεργες ποικιλίε, ξαφνικά δεν θα έχει δουλειά. Υπάρχουν τεράστιες ε, τράπεζες γενετικού υλικού σε όλη την Ευρώπη όπου προστίθενται νέες ποικιλίε κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι διαφορετικό από το θέμα της βιοπικιλότητας ε, που ε, εξαρτάται από το τι ζητάνε οι καταναλωτές. Είναι λοιπόν πολύ καλή η βάση που δημιουργήσε ο συνάδελφο και ελπίζουμε με κάποιες τροπολογίες να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο. προσβλέπω στη δουλειά αυτή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο, κύριο Στάδλερ και μετά Μάρτα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω εκεί όπως συνάδελφος Άγνιο σταμάτησε πιο πριν. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά αιτία, κανένας λόγος για αυτόν τον κανονισμό για τους σπόρους, για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και οι διαμαρτυρίες ε, των ανθρώπων ήταν ιδιαίτερα έντονες, ασυνήθιστα έντονες και σε ευρύτατο πλαίσιο. Πολλές αντιδράσεις είχαμε και το ανέφερε και η κυρία Κάνεμπαχ και στην Αυστρία οι πολίτες ε, με πολύ κριτικό τρόπο τοποθετήθηκαν και επικρίσεις. Είναι απόλυτα περίτη πρόταση που τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή την μανία ρυθμιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε μαζικές καλλιέργειες φυτικές εδώ που να εντάσσονται μέσα στα πλαίσια αυτά ή να έχουμε κάποιο είδους ανάγκες για να υπάρξει μια ρύθμιση σε σχέση με αυτά τα προϊόντα απλά και μόνο είναι τα συμφέροντα των αγροβιομηχανιών που θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι θέματα εχέγγυων και θέλω να υπενθυμίσω τα λόγια ε, που αναφέρθηκαν σε σχέση με τον κύριο Ντόρφμαν. Εκείνοι που αγοράζουν σήμερα φυτικό υλικό θα πρέπει να διασφαλίζονται ότι δεν ε, υπάρχει οπισθοδρόμηση να μην γνωρίζει τι πουλάει και τι αγοράζει. Δεν χρειάζεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ρυθμίσει ούτε κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η απώλεια εγγύηση πουθενά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να δικαιολογεί ένα τέτοιο κανονισμό. Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Εκείνοι που αγοράζουν φυτικά τέτοια προϊόντα μπορούν να συνεχίσουν να τα αποκτούν και να τα προμηθεύονται από άλλους γεωργούς. Και αν κάτι δεν πάει καλά μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει αποζημίωση. Δεν χρειάζεται με, με απόλυτη βεβαιότητα αυτός ο κανονισμός. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλυφθούν και άλλοι παραγωγοί με γραφειοκρατικές ε, ε, επιβαρύνσεις και με προσκόμματα και εμπόδια θα εξωθηθούν από την ε, αγορά. Διότι ποιοι είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν καλύτερα με γραφειοκρατική επιβάρυνση. Οι μεγάλοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις τα καταφέρνουν καλά. Οι μικροί δεν, δεν μπορούν να τα καταφέρουν και εξωθούνται από την αγορά. Και αυτό είναι επιζήμιο για τους μικρούς επιχειρηματίες. Έχουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν και ρόλο δεσπόζοντα στην αγορά έναντι πολύ μικρών άλλων. Αλλά ποιος πληρώνει πάντα, ο μικρός, ο μικρός, ο, κοινός θνητός σε σχέση με τις νης, τις ειδικέ γεωργικές πρακτικές διαχείρισης, πεδίο δραστηριοτήτων δηλαδή. Και εκεί ομοιογενείς παραγωγή και πιστοποιημένα προϊόντα πρέπει να μπορούν να εμπορεύονται από τους ε, ενδιαφερόμενους μέσα σε μια αλυσίδα, σε ένα πλαίσιο ας το πω έτσι αλληλουχίας που να διασφαλίζει τις ανάγκες τους. Και όχι να έχουμε εδώ τέτοιες υπερβολικές ρυθμίσεις. Υπάρχει αντίσταση των πολιτών μας κατά αυτής της μανίας ρυθμίσεων και διατάξεων. Συμφωνώ ε, και είναι πραγματικά περιττή αυτή η προσπάθεια όχι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω, δηλαδή να εξωθηθούν ακόμα περισσότερο οι μικρομεσαίοι από την αγορά και να έχουμε υποχρεωτική ένταξη όλων σε αυτές τις διατάξεις και ρυθμίσεις, το αντίθετο πρέπει να γίνει. Οι μεγάλοι πρέπει να εντάσσονται σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις, σε αυτούς να περιοριστούμε. Για τους υπόλοιπους που είναι μικρότερων διαστάσεων καλλιεργητής, καλλιεργητές δεν χρειάζονται κανονισμοί και προτάσεις της Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Στάλλερ, Μαρκ Ταραμπέλα και μετά Μισελ Μάρκ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πολλά υπάρχουν να πει κανεί για αυτό το κανονισμό που θέλει να αντικαταστήσει όλες τις οδηγίες. Είναι πολύ φιλόδοξο και φυσικά είναι εγωιτευτική αυτή η ιδέα της απλούστευσης που συχνά αναφέρεται. Πέραν αυτών όμως ε, τίθενται κάποια ανησυχητικά ζητήματα από το σχέδιο αυτό νομίζω. Και χωρίς να αρχίσω να αναφέρω μια σειρά άρθρων για να δώσουμε χρόνο για την ακρόαση που έχουμε αργότερα, δεν θα μιλήσω για το άρθρο 3 για την εμπορική διάθεση που ε, θέλει να αλλάξει ο κύριος ε, Σιλβέστρης, αλλά θα αναφερθώ σε τρία άρθρα. Το 36 αφορά τα υλικά εξειδικευμένων αγορών με μια τροποποίηση που κάνει ο κύριος συζητητής και που είναι μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι λίγο περιοριστικό, διότι γενικά, εντάξει δεν είμαι παρανοϊκός, αλλά έχουμε την εντύπωση δεδομένης της τεράστιας συγκέντρωσης ε, που μέσα στον χρόνο έχει γίνει στον κόσμο της εμπορικής διάθεσης και κυκλοφορίας διάδοσπορων, πόρων, είτε για τη γεωργία μεγάλων εκτάσεων, είτε για την αεραστεχνική κυπουρική, δηλαδή καλύπτει όλη τη, όλο το εύρος των θεμάτων ε, που επιτρέψει τους τη παρούσα Κομισιόν. Παρατηρούμε λοιπόν μέσα στον χρόνο αυτή τη συγκέντρωση και εμεί εδώ πρέπει να ακολουθούμε και τις λογικές που ακολουθούμε και σε άλλους τομείς ε, για την ανάπτυξη, για την οικονομία, για την ανάκαμψη, για την καταπολέμηση της ενεργείας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτός ο περιορισμός, αυτή η λέξη νη στο εξειδικευμένες αγοράς φαίνεται πολύ συμπαθητικό αλλά αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ελπίζουμε να αναπτυχθούν. Ιδίω επειδή οι καταναλωτές ζητούν αυτές τις ποικιλίε. Ε, όλο και περισσότερο τις περισσότερε παλιές ποικιλίε που επανέρχονται στη μόδα. Ε, Πώ να περιορίζουμε λοιπόν σε 10 υπαλλήλου και 2 εκατομμύρια τζίρο. Αν μετά από μερικά χρόνια βγάζουν 125, ωραία θα ε, καταπολεμηθεί η ανεργία σε περιοχές που το έχουν ανάγκη βέβαια. Αλλά λοιπόν αυτός ο περιορισμός δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει. Το άρθρο 57 αναφέρεται στις ποικιλίε, στις περιγραφές που αναγνωρίζονται επίσημα, μια περιγραφή που είναι πολύ δύσκολη και δύσκολη να υλοποιηθεί, αλλά μιλάμε για ποικιλίε που πρέπει να παράγονται στην περιοχή καταγωγής τους. Και εκεί βλέπω ένα περιορισμό. Ε, κάποιο προϊόν που φέρει το όνομα Κρυμαία, σπάνω δεν παράγεται μόνο στην Κρυμαία μπορώ να σας μιλήσω για πολλές ε, ποικιλίε που έχουν μεταφυτευτεί σε άλλες περιοχές ε, που έχουν ίσως την ίδια καταγωγή αλλά έδωσε μια ιδιαίτερη ποικιλία με εξελίξεις, διάφορες αλλαγές. Ε, αυτό οδηγεί και σε πλούτο, σε βιοποικιλία. Και αυτός είναι ένας περιορισμός λοιπόν που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά με αυτόν τον κανόνα είτε αναγκάζουμε τους μικρές επιχειρήσεις να έχουν ε, τις περιοχές όπου αναπτύσσεται το μέτρο ή εγκαταλείπουμε τη διατήρηση αυτών των ποικιλιών που με στο χρόνο έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν περάσει διάφορες ηλικίε. έχουν διαδοθεί σε διάφορες περιοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το άρθρο 57 θα πρέπει να ε, γίνει πιο χαλαρό και να τροποποιηθεί. Τώρα για να αναφερθώ στα άρθρα 135 και 136 όσον αφορά τα δικαιώματα καταχώρησης των ποικιλιών στους καταλόγους διότι εδώ δεν γίνεται καμία εξαίρεση για ποικιλίε που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Είναι οι πιο παλιές ε, ποικιλίε αυτές ε, από... Ε, σίγουρα υπάρχει κάποια επένδυση, αναμφίβολα, αλλά δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα δικαιώματα για φυτά που ε, κυκλοφόρησαν, που διαδόθηκαν μέσω κυπουρών, μέσω γεωργών, ε, υπάρχουν και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον. Έχω ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τον κατάλογο Βίλ Μωρά από τις αρχές του 20ου αιώνα και εκεί βλέπετε είναι 50, 60, 70 σελίδες ε, για τα ναρακά για παράδειγμα αλλά Σήμερα υπάρχουν 5-6 μόνο ήδη. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίβαρο ώστε να μπορούν όλοι να συνεπάρχουν, αλλά κυρίω επαναλαμβάνω οι ερασιτέχνε και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που, που μου ζητούν να αναπτυχθούν. Θα υποβάλω λοιπόν τροπολογίε ε, για αυτό το φάκελο που ελπίζω να σα βρω όλου σύμφωνου. Ε, ε, και ελπίζω λοιπόν ότι με, αν είμαστε στο διάλογο θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε αυτά. Δίνω το λόγο στον Μισελ Νταρντέν να, καλέσω την να, προσκα... να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία του Πανεπιστήμιου του Μπάρι με τον Πρίτανη τον Αντώνιο Ρίκιο. Μισελ Νταρντέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως μερικές φορές συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και μερικές εβδομάδες, το φάκελος αυτός δημιουργεί πάθη. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η εκστρατεία της οποίας είμαστε στόχοι όλοι. Είναι πολύ εύκολο να πατήσουμε ένα κουμπί για να πούμε την άποψή μας. Εγώ σας ομολογώ ότι προσωπικά δεν λαμβάνω υπόψη όλες αυτές τις εκστρατείες που κινητοποιούν τους βοηθούς μου όπως και τους βοηθούς των συναδέλφων. Εγώ δίνω περισσότερη προσοχή στον όσο, σε όσους έχουν το θάρρος να μου γράψουν. Σε αυτό το φάκελο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η συζήτηση για τον κόσμο της Γεωργίας ε, της γεωργικής παραγωγής έχει σχέση και με τα γεωργικά προϊόντα. Μιλάμε πολλές φορές για κλασικά προϊόντα, για προϊόντα εξειδικευμένων τα κτλ. Πιστεύω ότι η συζήτηση πρέπει να είναι η ίδια όσον αφορά και την παραγωγή του υλικού και την κυκλοφορία του υλικού και των σπόρων. Πρέπει αφενός να διασφαλίσουμε όλους τους γεωργούς που αγοράζοντας εμπορικά σπόρους χρειάζονται βεβαιότητα όσον αφορά την ομογένεια των παρτίδων, όσον αφορά τις υγειονομικές ε, ιδιότητες ε, και τις αντοχές που επισημαίνονται για τους εν λόγω πόρους. Ταυτόχρονα πρέπει να διαφυλάξουμε την ελευθερία του καθενός και ειδικότερα των ερασιτεχνών, την ελευθερία να χρησιμοποιούν τις ποικιλίε που επιθυμούν. Επίσης, σε σχέση με τα όσα είπα σήμερα το πρωί, πιστεύω ότι όλοι χρειαζόμαστε για το μέλλον διατήρηση της γενετικής πυκλομορφίας. Δεν πρέπει λοιπόν, ε, πιστεύω, να προχωρήσουμε σε μια, ένα νόμο ο οποίος θα σκοτώσει τον ένα για να προστατεύσει τον άλλο. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία η οποία θα επιτρέψει στους μεν να αναπτυχθούν διαφυλάσσοντας τους τους άλλους. Αλλά προσοχή στη συζήτηση μεταξύ μικρών και μεγάλων. Διότι ανοίγοντα την πόρτα στους μικρούς δεν κάνουμε κάτι. Ένας μπορεί να είναι μικρός έχοντας ένα προϊόν στο εμπόριο και να είναι μεγάλο στο παραγωγή αυτού του προϊόντο. Ή μπορεί κάποιο να είναι μικρό γιατί έχει πολλέ μικρές ποσότητες πολλών διαφορετικών προϊόντων. Ξεκινώντα κάποιο από μικρό μπορεί να γίνει μεγάλο. Έχει συμβεί. Ε, Κύριο Σιτσαρλατάνη γίνονται έτσι. Και πιστεύω ότι οι κανονισμοί αφήνοντα ε, ελευθερία στους μικρούς ε, θα πρέπει να παρέχουν μια ελάχιστη ποσότητα ασφάλειας ώστε αύριο να υπάρχει περιθώριο ή υπό την ευρωπαϊκή σφραγίδα για οποιοδήποτε οικονομικό βανδαλισμό. Πολύ ωραία συνάδελφοι. Ε, ευχαριστούμε για όλες τις ε, παρεμβάσεις. Δείξαμε ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία για ένα θέμα στο οποίο πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σέτζοφ Σιλβέστρη. Ε, προετοίμασε μια καλή βάση για συζήτηση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Έρικ Μουτλέρ. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον Σέτζο Σιλβέστρης για να απαντήσει στα σχόλια που ακούσαμε. Παρακαλώ κύριε Μουτλέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό πράγματι δημιουργεί πάθη και ήθελα να επιβεβαιώσω μπροστά σας τόσο έχω ήδη πει. Όταν γράψαμε αυτό το σχέδιο, αυτό που σκεφτόμασταν ήταν φυσικά απλούστευση των γνωστών 12 οδηγιών, στις οποίες αναφερθήκατε ορισμένοι, αλλά κυρίως αυτό που είχαμε στο νου μας ήταν να αυξήσουμε την ευελιξία των πιστοποιήσεων και να ενθαρρύνουμε την κοπικιλότητα. Πολλοί από εσά το είπατε κυρίως όσον αφορά αυτές τις μικρές ε, ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η τις μεγαλες επιχειρησεις επιθυμια μας ήταν οι μικροεπιχειρήσεις αυτές ε, που κυκλοφορούν στην αγορά σπόρους ε, ποικιλιών με λίγους υπαλλήλους μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να μην εξαφανιστούν λόγω του ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς θέλησαμε επίσης να ενθαρρύνουμε την τοπική παραγωγή τις μικρές ε, περιορισμένες αγορές ε, για αυτό το λόγο. Εξαιρέσαμε από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού τις ε, δωρεάν ανταλλαγές μεταξύ ατόμων. Εδώ είχαμε ως στόχο φυσικά τους γεωργούς που μπορούν να ανταλλάσσουν σπόρους αλλά και τους ερασιτέχνες των... της Κυπουρικής που ανταλλάσσουν σπόρους για λουλούδια για παράδειγμα. Θέλαμε να προστατέψουμε αυτό την τεράστια γενετική κληρονομιά. Δεν θέλαμε ένα κατάλογο ειδών ε, με μειωμένο αριθμό ποικιλιών καθόλου. Κανείς εδώ δεν θέλει να μειώσει τη βιοποικιλότητα. και σίγουρα όχι η Κομισιόν. Διότι μάλιστα είτε μιλάμε με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας είτε Περιβάλλοντος, ενθαρρύνουμε όλη τη βιολογική γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τα προς εξαφάνιση ήδη τα είδη που από εξαφάνιση. Θέλαμε λοιπόν να προσφέρουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα παρέχει πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα σε αυτές τις ε, εξειδικευμένες αγορές, σε αυτές τις παλιές ε, ποικιλίε. Συμφωνούμε με τα όσα είπαν ο κ. Γιάννη και ο κ. Σοφμαν ότι ανεξαρτήτως του μεγέθους επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, αυτές θα πρέπει να παράσχουν στους αγοραστές των σπόρων τους, είτε πρόκειται για επαγγελματίες αγρότες, είτε πρόκειται για ερασιτέχνες, θα πρέπει να προσφέρουν σπόρους υψηλής ποιότητας που να αντιστοιχούν πραγματικά στις επιλογές του καταναλωτή. Ώστε όποιος αγοράζει τους σπόρους αυτούς ε, ή τους, ε, τους σπόρους ε, δέντρων να μην βρεθεί μερικά χρόνια μετά ή στο τέλος της σεζόν με προϊόντα που δεν επιθυμούσα. Αντιθέτω, αυτό σε διαφορετικό πλαίσιο θελήσαμε για αυτέ τι μικροεπιχειρήσει των λίγο κάτω των 10 υπαλλήλων να τι εξαιρέσουμε από την υποχρέωση επιθεωρήσεων από τι αρχέ. Διότι φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα πιστοποίηση απαιτούν την παρέμβαση των αρχών των κρατομελών. Και αυτέ οι παρεμβάσει πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Έτσι προτείναμε σε ένα άλλο κείμενο, στο κείμενο περιελέγχων, την εξαίρεση των υποχρώσεων αυτών ε, για τις μικροεπιχειρήσεις. Ήθελα επίσης να επιμείνω ότι στο κείμενο αυτό προσφέρεται ένα νέο νομικό πλαίσιο για την εμπορική διάθεση των σπόρων. Αλλά επιμένω πρέπει να δείτε τις εξαιρέσεις του άρθρου 1. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι μπορεί να κατευνάσει πολλές ανησυχίες, πολλά προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα. Ο κύριος Λάιον αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του τομέα των σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας αυτός ε, είναι παγκόσμιος ε, ε, κυρίαρχος, είναι ηγέτης στην πρώτη θέση. Η Ευρώπη εξάγει σπόρους σε ολόκληρο τον κόσμο, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή ομάδα χωρών στον κόσμο και αυτό χάρη στην ποιότητα και τη σοβαρότητα των επιχειρήσεων που κυκλοφορούν στην αγορά διεθνώ, στη διεθνή αγορά στους σπόρους. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και οι μικρές ε, περιφερειακές ή εθνικές επιχειρήσεις προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Σκέφτομαι τον Αρακά που ανέφερε ο κ. Σταραμπέλα, ε, μπορεί να εξαφανίστηκαν από τον κατάλογο του Βιλμορά, ίσως διότι κανείς πια δεν ε, αγοράζει. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ ε, ψαγμένων, ας πούμε, ραστεχνών οι οποίοι έχουν συμβουληθεί τέτοιους καταλόγους και όχι μόνο τους επίσημους καταλόγους. Στόχος επίσης αυτού του κανονισμού είναι να οδηγήσει σε μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματιών αριστεχνών, μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις, πολλά πάθη, πολλά χρήματα. Ωστόσο αυτή η ισορροπία, όπως πενθύμισε ο κ. Ντάντα, είναι σημαντική θα τελειώσω με τρία νούμερα. 70% των επιχειρήσεων που διαθέτουν σπόρους στην αγορά για λαχανικά είναι μικροεπιχειρήσεις. 80% των επιχειρήσεων που κυκλοφορούν στην αγορά καλοπιστικά φυτά είναι μικροεπιχειρήσεις. Και 90% των επιχειρήσεων που κυκλοφορούν στην αγορά ε, κλίματα είναι μικροεπιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο τομέας αυτός δεν ε, ε, έχει απορροφηθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες στιγματίζουμε βέβαια αλλά κυριαρχείται από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και στόχος του κανονισμού αυτού ήταν να τους παρασχεθεί ένα νομικό πλαίσιο ώστε αυτές με απόλυτη νομική βεβαιότητα και ασφάλεια να μπορούν να λειτουργήσουν προσφέροντας ε, βεβαιότητα στους καταναλωτές, εραστέχνες ή επαγγελματίες, ό,τι αγοράζουν, σπόρους που αντιστοιχούν σε αυτό που αναφέρεται στον κατάλογο. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε στην παρούσα φάση και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε με τον κύριο Σιλβέστρη, τον κύριο Σιγητή και τους κύριους συγητές με σκόχο τη βελτίωση του κειμένου αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Σιλβέστρης ώστε να απαντήσει στις πολλές ερωτήσεις που ακούσαμε, Σέρτζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και ευχαριστώ για τις προτάσεις τους, για την προσοχή που έδωσαν στη συζήτηση που διεξάγουμε εδώ. Ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την ε, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου του Μπάρι με τον εκπληκτικό ε, Πρίτανη Εγώ έχω πάρει το πτυχίο μου, οπότε πλέον δεν τον φοβάμαι. Τον γνώριζα τον κύριο Πρέιταν αυτό και πρόκειται για εξαιρετική σύμπτωση. Θα ήθελα να καθισχάσω ορισμένου συναδέλφου, ειδικότερα τον συνάδελφο Άγνιο και Στάντλερ. Δεν αποφάσισα εγώ, ούτε αποφασίσαμε εμεί να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή ο κανονισμό αυτό. Το ανέφεραν και ο συνάδελφο κύριο Άγνιου και ο συνάδελφο κύριο Στάντλερ. Σίγουρα δεν ήταν η καταλληλότερη στιγμή δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να επανεξετάσουμε τους κανόνες για την αγορά του σπόρων και του πολυπλασιαστικού υλικού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους με τη σειρά. Στον συναδέλφο Οσλεγγ θα ήθελα να πω εκτιμώ πραγματικά τις προτάσεις σας και τη διάθεσή σας για συνεργασία Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ε, για ε, το σχέδιο αυτό. Είπε σαφώ ε, ο Σνάλ δεν ζητάμε προνόμια για του παραγωγού, αλλά ούτε θέλουμε να περιορίσουμε αυτό τη δυνατότητα. Σίγουρα αυτή είναι η λογική βάση τη οποία πρέπει να κινηθούμε, αλλά εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται ρύθμιση για τη διατήρηση των κεκτημένων. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κύριος Ντόρφμαν είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Συχνά οι αγοραστές ε, στρέφονται στην πλησιέστερη αγορά, κυρίως για τα φυτά, όχι τόσο πολύ για τους πόρους. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις και αυτές ορίζονται ε, επιχειρήσεις εξειδικευμένων αγορών θα υπάρχει στην αγορά μη ελεγμένο, μη πιστοποιημένο υλικό που θα προέρχεται παρόλα αυτά από μικρές επιχειρήσεις και θα καθορίζει παραγωγές μεγάλων σημαντικών ε, εκτάσεων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταφέρουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία ώστε να εγγυόμαστε ότι τόσο η εξειδικευμένη αγορά και η σχετική παραγωγή δεν θα υφίστανται γραφειοκρατία την οποία κανένας δεν επιθυμεί, ούτε εγώ να υπάρχει τέτοιο μονοπόλιο μόνο για μεγάλους παραγωγούς αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τους αγοραστές, τους καταναλωτές. Ήθελα να φέρω ένα στοιχείο που μου φαίνεται ότι προκύπτει από αυτή τη συζήτηση και που εκτιμώ ιδιαίτερα. Σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, συμφωνούμε στο εξή. Ο ορισμός της εξειδικευμένης αγοράς δεν μπορεί να σχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης. Και γιατί αυτό, και θέλω να το πω καθαρά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδος κερδοσκοπίας. Εάν οριστεί εξειδικευμένη αγορά βάσει του μεγέθους της επιχείρησης με ένα νότατο όριο των 2 εκατομμύριων ευρώ όπως ε, προτείνει η Κομισιόν, που μπορεί να μας κάνει να να πούμε γιατί όχι ένα 9 εκατομμύρια για παράδειγμα. Τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση, κάτι πολύ απλό ότι ορισμένες επιχειρήσεις για να αποφύγουν να υπόκεινται στις διατάξεις του παροντός κανονισμού καθώς θα αναπτύσσονται με τα χρόνια και θα ξεπερνούν τα δύο αυτά εκατομμύρια, το όριο δηλαδή για την ένταξη στον ορισμό των ε, παραγωγών ε, ε, εξειδικευμένης αγοράς χωρίζονται σε δύο επιχειρήσεις και συνεχίζουν να μην υπόκεινται στον κανονισμό αυτούς και κινδύνους πρέπει να, φύγουμε, να αποφύγουμε αλλά θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι Και να υπενθυμίσω, ο συνάδελφος Όσβινγκ είπε πολύ σωστά, πρέπει να βρούμε έναν ορισμό σωστό, ισορροπημένο. Καινούριο όμως, όχι αυτόν της Κομισιόν. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Κάδεμπαχ. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε νέα γραφειοκρατία. Πρέπει να διαφυλάξουμε όμως και τη βιοπικιλότητα. αυτή διαφυλαστεί κυρίως από τους καταναλωτές όπως πολύ σωστά είπε κάποιος διότι οι παραγωγές βασίζονται στις απαιτήσει της αγοράς, στη ζήτηση της αγοράς που κατά την απόψή μου είναι ο πρώτος υπερασπιστής της βιοπικιλότητας. Ε, σκέφτηκα όλες αυτές τις τροπολογίες που είπε η κυρία Κάδεμπαχο, θα προτείνει, θα τις μελετήσω και με τους κυρίωδεις συζητητές και θα τις εξετάσουμε με πνεύμα συνεργασίας. Επιφυλασσόμαι να σας στείλω συγκεκριμένες απαντήσεις ε, με την πρόταση της Κομισιόν και το σχέδιο έκθεσης διότι είπε η κυρία Ρόντου το ότι εάν οι απαντήσεις σας είναι πλήρες δεν θα υποβάλω τροπολογίες. Οπότε θα προσπαθήσω να σας στείλω ακριβείς απαντήσεις ώστε να μειώσω και τη δική σας δουλειά και την δική μας δουλειά στην Επιτροπή ε, της Αλλά να σας πω κάτι, όσον αφορά το υλικό των εξειδικευμένων αγορών, θα πρέπει να ορίσουμε τις εξειδικευμένες αγορές βάσει άλλων στοιχείων, ε, αφήνοντας την Κομισιόν μέσω της πράξεων να ορίσει τις ποσότητες και με τοπικές παραγωγές φυσικά με δυνατότητες εμπορικής διάθεσης ε, αρκετά ελεύθερης. Με τις τροποποιήσεις μου είναι δυνατόν το νέο φυτικό υλικό να διατεθεί στην αγορά. Για τις παλιές ε, ποικιλίε του αρθρό 57 προβλέπει με μια ελαφριά καταχώρηση να κυκλοφορούν στην αγορά παραδοσιακές ποικιλίε. Εγώ θεωρώ ότι το άρθρο αυτό βοηθά στη διατήρηση τη κυκλοφορία ε, στην αγορά των προϊόντων αυτών και τη βιοπικιλότητα. Αυτή η έκθεση όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα υλικά δεν προβλέπει κάτι. Όσον αφορά την ασφάλεια, αυτό είναι από τα κέρια σημεία τη έκθεση. Το έχω γράψει. Θεωρώ ότι ο κανονισμό αυτό θα πρέπει να παράσχει και εγγυήσει και για τους αγοραστές και όχι μόνο πρότυπα για τους παραγωγούς. Με τον συνάδελφο Ντόρφμαν τον ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, ε, για τις υποδείξεις που έκανε και σίγουρα συμμερίζομαι και τα όσα είπε ο συνάδελφος κ. Γιάρα. Εγώ δεν μίλησα για περιφερειακές αγορές, αλλά για τοπικές αγορές στην εκθεσή μου. Ο ορισμός της τοπικής αγοράς δεν έχει μπει ακόμα στην έκθεση, αλλά πιστεύω ότι και... Πιστεύω ότι η συζήτηση που θα κάνουμε συνέχεια θα μας βοηθήσει να ορίσουμε καλύτερα το καθεστώ αυτού του τύπου. Την προσέγγιση μάλλον αυτού του τύπου, εφόσον συμφωνήσουμε εντό τη επιτροπή αυτή. Ο συνάδελφο Γιάρα ε, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα το οποίο και εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα. Είπε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση, να έχουμε ένα σαφή ορισμό μεταξύ του επαγγελματία και του μη επαγγελματία να υπενθυμίσω στον φίλο Πίτερ ότι για την ε, ΠΑΚ χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να καταλάβουμε ποιοι ήταν επαγγελματίε και ποιοι όχι. Και τέλος είπαμε ουσιαστικά στα κράτη-μέλη αποφασίστε εσείς. Εάν καταφέραμε με αυτή την έκθεση να καταλήξουμε, τουλάχιστον για αυτή την έκθεση να ορίσουμε ποιοι είναι επαγγελματίες φορείς και ποιοι όχι, πιστεύω ότι θα έχουμε καταφέρει ένα μικρό θαύμα διότι επί του ίδιου θέματος, συζητώντας την κοινή αγροτική πολιτική, καταφέραμε μόνο να πούμε ποιος είναι ενεργός ε, γεωργός, αλλά μετά είπαμε στα κρατημέλη πρέπει να βρείτε εσείς μια λύση. Ναι, οι δυσκολίες για τα φρούτα είναι κάτι που πρέπει να εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ τον Πίτερ που το υπογράμμισε. Με τον συναδέλφο Λάιον πιστεύω ότι λειτουργούμε στο ίδιο πνεύμα και θα πρέπει να προχωρήσουμε επιδιώκοντας να βρούμε μια σωστή ισορροπία ώστε να αποφύγουμε οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό αυτόν για να αποφεύγουν να καταχωρούν μια ποικιλία αλλά θα πρέπει επίση να βοηθήσουμε να εξασφαλίζεται η βιοπικιλότητα και οι εξειδικευμένε αγορές χωρίς η γραφειοκρατία να περιπλέξει περισσότερο την εργασία των μικρών παραγωγών Συνάδελφε Τραμπέλα ε, κάνατε τέσσερι ερωτήσει, αναφέρετε τέσσερα προβλήματα για τέσσερα άρθρα του κανονισμού, τα άρθρα 36, 57, 135 και 136. Εγώ αυτά τα τέσσερα νούμερα θα τα παίξω στο λότο την επόμενη εβδομάδα και σας υπόσχομαι ότι θα μοιραστούμε τα κέρδη με τον συναδέλφο Ταραμπέλα. Αυτά τα τέσσερα άρθρα είναι τα άρθρα πυρήνε του κανονισμού. Είναι πολύ σημαντικά για τη δεξιδικευμένη αγορά. Έχουμε συζητήσει πολύ, είναι κάτι που μα ανησυχεί. Πρέπει να εμβαθύνουμε για τον ορισμό αυτόν. Τώρα όσον αφορά τον ορισμό της εμπορικής διάθεσης των ποικιλιών που παράγονται στην περιοχή καταγωγής. Σίγουρα, προφανώς, δεν μπορούμε να περιορίσουμε την εμπορική διάθεση στην περιοχή καταγωγής. Αυτή, το παράδειγμα της ντομάτας Κρεμαίας ε, ήταν πολύ χαρακτηριστική. Πολύ χαρακτηριστικό για τα άρθρα 135-136. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτό κάποια στιγμή αφού το μελετήσω. Πιστεύω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα επικοδομητική με τον συνάδελφο Νταντέν, ε, το είπα και προηγουμένως. Συμμερίζομαι αυτή την ιδέα ότι αυτός ο ορισμός εξειδικευμένης αγοράς ε, που σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, να δημιουργήσει παράνομους μηχανισμούς ε, αποφυγής των περιορισμών αυτών. Δεν πρέπει εμείς να δώσουμε τέτοια κίνητρα. Αυτές τις δύο έννοιε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την άποψη των αγοραστών και των καταναλωτών. Την ιδέα ότι ο κανονισμός αυτός πρέπει να θεωρείται απαραίτητος όχι γιατί έχει μια μανία αριθμίσεων των πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να διαβεβαιώσουμε τους αγοραστές ότι μπορούν με την ισχύ τους να αγοράζουν ήδη τα οποία αντιστοιχούν στις περιγραφές είναι υγιή και δεν μεταφέρουν ε, νόσους των φυτών. Αυτή είναι η στόχη. Από την άλλη Στόχος μας πρέπει να είναι να μην αυξήσουμε τον διοικητικό φόρτο και κυρίως για τους μικρούς παραγωγούς που σίγουρα εμπλουτίζουν την αγορά και πρέπει να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται διότι δεν θέλουμε μονοπόλια στις αγορές αυτές των φυτών. Εάν έχουμε αυτά τα δύο σημεία αναφοράς καθαρά στο μυαλό μας, ο στόχο θα μπορέσουμε να εργαστούμε βρίσκοντας σωστά ισορροπίες στη δομή και στους ορισμούς ε, του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη δραστηρία και επικοδομητική του συμμετοχή, για τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Ε, θα στείλω κάποιες παρατηρήσεις στην κυρία Ρόντου, στο όπως υποσχέθηκα, και θεωρώ ότι αν κρατήσουμε αυτή την οδό μια προσέγγιση μη ιδεολογική, αλλά υποβάλουμε προτάσεις όλοι, έχοντας σαφείς τους στόχους στο μυαλό μας, ε, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε γρήγορα να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη στιγμή για τέτοιες αντιφατικές ε, συνομιλίες, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα του Κοινοβουλίου μέσω ενός κειμένου, μέσω της εκπόνησης ενός κειμένου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού, στο οποίο ευθυνόμαστε. Ευχαριστώ όλους. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστρη, ευχαριστούμε την Κομισιόν και όσους, όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, πριν δώσουμε... Ξεκινήσουμε την ακρόασή μας ε, με τους έξι εμπειρογνώμονες που αναμένουν. Χρειαζόμαστε μερικά λεπτά για το σημείο 14, το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μέτρα προστασίας κατά των επιζήμενων οργανισμών για τα Υπερβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Ε, δίνω τον λόγο στον κύριο Φαϊμόν ε, για αυτό το τελευταίο σημείο και παρακαλώ να συντομεύουμε για να μην υπάρχουν προβλήματα με την ακρόαση. Ευχαριστώ. Κύριε Φαϊμόν. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Μετά από μια σε βάθος προσεκτική ανάγνωση αυτής της πρότασης και διαβούλευση με τους σκιώδεις εισηγητές και τους πραγματογνώμενους και παίοντε σε αυτό το τομέα, και καθηγητές και επιστήμονες ε, η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ορθολογική. Ο εξυγχρονισμό τη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική υπόθεση, λαμβάνοντα υπόψη του αυξημένου κινδύνου. Είναι επίση θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω πακέτο μέτρων υποβάλλει αυτή την πρόταση, που εμπεριέχει όλη την αλυσίδα για τα τρόφιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων όμω που πρέπει να εξεταστεί από πλευρά μα. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό γεωγραφικά το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας να το περιορίσουμε και να αποκλειστούν κάποιες περιφέρειες. Η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια κοινή επικράτεια. Σε αυτή την επικράτεια πρέπει κοινοί κανόνες να ισχύουν. Δεν είναι σωστό κάποιοι κανόνες να ισχύουν μόνο σε ένα μέρος της επικράτειας, κάποιοι άλλοι να ισχύουν για άλλες περιφέρειες. Κάτι τέτοιο δημιουργεί προσκόμματα και εμπόδια και δεν, θα ανταποκρινόταν στη σωστή μεταχείριση της ενιαίας επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι δεν συνδέεται επαρκώς με διεθνείς προδιαγραφές αυτή η πρόταση που η κοινοβουλευτική μας επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την πτυχή και πιστεύω ότι όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει στο σύστημα των προστατευτικών μέτρων να μπορούν να ενταχθούν έναντι των επιζήμιων για τα φυτά ασθενειών. Θεωρώ ότι πρέπει να καταπολεμηθούν τα παράσιτα και μάλιστα να υπάρχουν δυνατότητες να γίνει αυτό και σε δημόσιες εκτάσεις. Θεωρώ ότι πρέπει ένα μεγάλο πλαίσιο διαφάνειας να δημιουργηθεί. Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε οποιασδήποτε απώλειες. Οι κάτοχοι, οι ιδιοκτήτες, εκείνοι που έχουν την κυριότητα ε, τέτοιων ε, εκτάσεων πρέπει έγκαιρα να ειδοποιούνται και να ενημερώνονται. Και σε σχέση με το ότι το νέο σύστημα ε, θα οδηγεί στην αντιμετώπιση των επιζήμιων για τα φυτά ασθενειών με μια υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιτευχθεί συγκρίσιμη με εκείνη την υποστήριξη και ενίσχυση όπως ισχύει στον, κτηνοτροφικό, στον ε, κτηνιατρικό τομέα. Και σε σχέση με την ε, διάρκεια 2014-2020, η διάρκεια αυτή είναι σωστή και αναγκαία. Είναι ένα αναγκαίο βήμα αυτό που πρέπει να γίνει. Από πλευράς ε, εισηγητού θεωρείται ότι τα μέτρα αυτά υπερβολικά πολλές δραστηριότητες μεταθέτουν και ε, αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη πολλά καθήκοντα και υποχρεώσεις θα επομισθούν. Για παράδειγμα υπερβολική υποβολή εκθέσεων και στοιχείων από πλευρά συγητού ε, θεωρείται ότι πολλά πράγματα τα οποία μπόρεσαν και ήταν δυνατόν να ρυθμιστούν σε συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών, σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινηθούμε και όχι να μετατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα θέματα θα μπορούν με τροπολογίες, ε, τροποποιήσεις ε, να διευθετούνται. Έχω καταθέσει 30 τόσες τροπολογίες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το πεδίο και ισχύσε. Θα ήταν σημαντικό να μπορέσει να ισχύσει αυτό το πακέτο. Ταυτόχρονα και οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί εθνικά αρμόδιοι να έχουν αρκετό χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους να προσαρμοστούν. Αυτό θα απαιτήσει δύο ή τρία χρόνια. Οι δικοί μου επαΐοντες με τους οποίους συζήτησα ισχυρίζονται από πλευρά της χώρας μου ότι τουλάχιστον δύο χρόνια θα απαιτηθούν για αυτές τις προσαρμογές. Όταν αυτό το νομοθέτημα θα αρχίσει να ισχύει το 2015 θα απαιτηθούν λοιπόν, θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι το 2018 αναφέρει ο Μιλτής ως ε, ημερομηνία ε, ενημερώθηκα ότι 65 τροπολογίες έχουν κατατρεθεί σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Molto bene, grazie collega Fimont, grazie anche per la rapidità con cui ha fatto la sua esposizione. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Φαϊμόν. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε τόσο γρήγορα την ε, παρουσίαση ε, της εκθεσής σας. Η Κομισιόν θέλει κάτι να προσθέσει. Παρακαλώ. Ωραία Θαμόρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Η σκιώδηση συγχύτρια που δεν μπορεί να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και σε σχέση με τις εκλογές στην Ονδούρα έπρεπε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πολύ σύντομα να διαβιβάσω την τοποθέτησή της για αυτή την έκθεση. Πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε για αυτή την έκθεση, τη σύνταξή της. Οι κυριότερες ιδέες μας είναι οι εξής. Είναι αναγκαίο να εισαχθεί στον θεμελιώδη κανονισμό ένας κατάλογος αυτών των ασθενειών και να υπάρξει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ως σημαντικό στοιχείο αυτού του νομοθετικού πακέτου. Επίσης, να να έχουμε περιορισμό, να έχουμε καθορισμό των προστατευόμενων ζωνών σε σχέση με τις ασθένειες αυτές ώστε να αποφύγουμε αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την εμπορία κάποιων προϊόντων. Είμαστε υπέρ του ότι οι εισαγωγέ προϊόντων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από χώρε που έχουν τι άδειε ε, και ε, να υπάρχει προσαρμογή στα όσα απαιτούνται από, την κτηνοτροφική, από τον κτηνοτροφικό κανονισμό. Αυτό απαιτεί μια ριζική αλλαγή νοοτροπία, διότι αυτή τη στιγμή γενικά επιτρέπονται οι εισαγωγέ ε, και μόνο αν υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αυτά είχα να πω ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ντάντσιλα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς αυτή η νομοθετική πρόταση στόχο έχει να ενισχύσει ε, τα μέτρα πρόληψης ε, και τα μέτρα έγκαιρης αντίδρασης ε, σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων επιβλαβών οργανισμών. Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργήσουμε και να βρούμε τις πιο κατάλληλες λύσεις καταπολέμησης όλων των παραγόντων που έχουν αρνητικές ε, συνέπειες ε, στην γεωργία, το σύνολο της ε, τροφικής αλυσίδας και τον γεωργικό τομέα, ώστε να εκριζώσουμε αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε μέτρα πρόληψης που μπορούν να λάβουν οι γεωργοί για να ελαχιστοποιήσουν τον ε, κίνδυνο εμφάνισης ε, των ε, επιβλαβών οργανισμών προτού εφαρμόσουμε πιο ριζικά μέτρα όπως είναι η χρήση των φυτοφαρμάκων. Η υγεία των φυτών είναι απαραίτητη για τη γεωργία και για την ανάπτυξη των δασών και είναι επίσης σημαντική για την προστασία της βιοπικιλότητας και την προστασία του οικοσυστήματος όλα τα θέματα που συνδέονται με τους επιβλαβείς οργανισμούς των φυτών ε, θα πρέπει να τα δούμε ε, ε, όχι μόνο από την οικονομική πλευρά αλλά πρέπει να εξετάσουμε και την προστασία του συνόλου της ε, διατροφικής αλυσίδας. Η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης απειλείται και σύμφωνα με τις στατιστικές των τελευταίων ετών θέματα υγείας των, ε, προβλήματα υγείας των φυτών έχουν αυξηθεί ε, στην Ευρώπη, ε, αποτελούν το εμπόριο και η αλλαγή του κλίματος. Τα μέτρα με στόχο τον έλεγχο των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών θα πρέπει να ληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της ε, πρόληψης για να προστατεύσουμε την ε, επιστητική ε, ασφάλεια και το περιβάλλον. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, να παρέχουμε χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οπτική και κατά την υποβολή ε, τροπολογιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το σύνολο της ε, ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι θα εξετάσουμε το θέμα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο θέμα αυτό, διότι η κατεξουδότηση πράξη δίνουν υπερβολικά πολλή εξουσία στην Κομισιόν και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε την κυρία Ντάντσιλα. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καναλών, Ερικ Μοντιλέ, να μας κάνουν μερικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Φαϊμόν. Με ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, αν θέλετε, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Να πω δύο λόγια για τα προβλήματα των περιφερειακών περιοχών, των άκρως απομακρυσμένων περιοχών στις τροπικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμάς. Για εμάς οι ζώνες αυτές ε, ανάλογα με το κλίμα, τα φυτά, ε, τις ε, τοπικές συνθήκες έχουν ιδιαιτερότητες που μας οδηγούν στο να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για περιοχές διαφορετικές από την υπηρετική επικράτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προτείνουμε η σημερινή κατάσταση όπου δεν υπάρχει ελεύθερη συναλλαγές μεταξύ της Υπήρου και των άκρως απομακρυσμένων αυτών περιοχών να ρυθμιστεί ώστε να μην εισαχθούν ε, στην Ευρώπη ασθένειες που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί λόγω της κλιματικής αναλλαγής. Επίσης όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τη σχετική λίστα εμείς επιθυμούμε να υπάρχει κάποια ευελιξία να μπορούμε να τροποποιήσουμε τη λίστα αυτή σε συνάρτηση με νέου επιβλαβεί οργανισμού που ενδεχομένω θα εμφανιστούν στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτών των προβλημάτων εισαγωγών. Επιθυμούμε λοιπόν η λίστα αυτή να μην ε, είναι παγιωμένη, να μπορεί να τροποποιηθεί. Δύο λόγια για τις χρηματικές αποζημιώσεις για τους γεωργούς θεωρούμε ότι σίγουρα είναι ωφέλιμο για τη γρήγορη και μαζική εκρίζωση σε περίπτωση εμφανισής νέας Είναι σημαντικό λοιπόν οι γεωργοί να μπορούν να λάβουν αποζημιώσεις ε, όταν τους υποχρεώνουμε να κόψουν δέντρα, να καταστρέψουν καλλιέργειες. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για οπροφόρα δέντρα τα οποία χρειάζονται 5 με 10 χρόνια μέχρι να αποδώσουν προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να προβλέψουμε μια τέτοια οικονομική αποζημίωση. Η εισαγωγή φυτών από τρίτες χώρες ε, αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό ζήτημα που μας ανησυχεί. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε πολλά παραδείγματα τα πιο πρόσφατα είναι οι ασθένειε για τις ελιές στην Πουλιά, στο νότο της Ιταλίας. Επίσης είχαμε ίου στα πορτοκαλιά στη Σικελία. Είχαμε την όσο για τα σφήνικες ε, στη Μεσόγειο εδώ και μια δεκαριά χρόνια. Πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εισαγωγές αυτές. Δεν μιλάμε για αύξηση της γραφειοκρατίας. Μιλάμε για την προστασία πολύ απλά των γεωργών, των καλλιεργιών μας, των καλοπιστικών μας φυτών. Θεωρούμε ότι οι εισαγωγές ε, αυτές ε, ενέχουν κινδύνους ενδεχομένους, αλλά μπορούμε να τους διαχειριστούμε ή να τους απαλείψουμε. Αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο προποθέτει και συνεπάγεται κάποιες απαιτήσει, αναλύσεις, εργαστηριακές, ε, δοκιμές και δεν μπορεί να θεωρείται διοικητικό φόρτο. Ε, αυτά είναι τα σχολεία μα στην παρούσα φάση. Ωραία, ευχαριστούμε τη Γενική Διεύθυνση Υγεία. Ε, τον λόγο στον κύριο Φαϊμόν για να ολοκληρώσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι την 6η Δεκεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών. Και ευελπιστώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε αίσιο πέρασα για αυτή την έκθεση. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε και θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε και ζητώ συγγνώμη από τους εμπειρογνωμονές μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση μας για την υγεία των φυτών. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως. Έχουμε έξι σημαντικούς εμπειρογνώμονες. Ξεκινάμε με την κυρία Κρίστιν Κιάγκο, διευθύντρια της ε, Υπηρεσίας Προστασίας της Λετωνίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και ταυτόχρονα να ζητήσω από τον συναδέλφο κύριο Σιλβέστρους αν θα μπορούσε να έρθει στην έδρα της Προεδρίας. Ευχαριστώ. Lies paldies, godātie deputāti, dāmas un kungi. Jā, es esmu Kristīna Kjāgo, valsts auga aizsardzības dienesta direktora. Κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Λέγομαι Κριστίν Κιάγκο. Είμαι διευθυντής της Κρατικής Υπηρεσίας Προστασίας των Φυτών της Λετωνίας και ασχολούμαι με την εφαρμογή της νομοθεσίας. και με την δημιουργία νέας νομοθεσίας. Μπορώ λοιπόν να σας μιλήσω ε, εκ μέρους των γεωργών μας και των επιρρογνωμόνων μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, ε, για την εκπόνηση δηλαδή αυτού του εγκώδους εγγράφου, ε, που προσπαθεί να εναρμονίσει τα θέματα υγείας των φυτών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Στην πρώτη διαφάνεια λοιπόν βλέπετε κάποιες γενικές πληροφορίες. Η, η υγεία των φυτών δεν είναι λιγότερο σημαντική από την διατροφική ασφάλεια, ε, θέματα κτηνοτροφικά και η, ε, η υγεία των φυτών δεν είναι απλά οικονομικό θέμα. Έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με την ε, εξέλιξη του κράτους, ε, τι μέλλον θα έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ξέρουμε ότι το κλίμα αλλάζει και αυτό επηρεάζει την υγεία των φυτών. Ε, ο κόσμος συνήθως δεν ε, θυμάται ε, το παρελθόν, το μακρινό παρελθόν ε, και η υγεία των φυτών είναι σαν ένα θετό παιδί. Βλέπουμε ότι οι συνέπειες θεμάτων υγείας των φυτών είναι πολύ σημαντικές. Ε, υπάρχουν προκλήσεις που μπορούν να ε, επηρεάσουν ε, διάφορους τομείς όπως είναι η δασοκομεία. Όσον αφορά λοιπόν αυτόν τον κανονισμό, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλοι ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον IPPC, που Υπάρχουν λοιπόν θέματα ορολογίας και του, το, πώς έχει μεταφερθεί στον κανονισμό αυτή η σύμβαση. Ε, έχουμε για παράδειγμα τον ορισμό των ε, νέων οργανισμών. Σε χώρες με καλά ε, φυτογενομικά πρότυπα ε, δεν θα αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα. Επίσης έχουμε ε, το θέμα των διαφόρων ε, ειδών. Για παράδειγμα, ο κανονισμός δεν αναφέρεται σε ζυζάνια. Ο τομέας αυτός λοιπόν θα ρυθμιστεί ε, στην νομοθεσία για το περιβάλλον, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα διότι θα ε, απαιτηθούν περισσότεροι πόροι. Οι εμπορικοί μας εταίροι γνωρίζουν ότι υπάρχουν ζυζάνια και οργανισμοί καραντίνας και στον κανονισμό υπάρχει σχετική ρύθμιση, δημιουργούνται όμως νέα συστήματα, νέοι νόμοι Όλα αυτά όμως απαιτούν περισσότερη χρηματοδότηση. Αυτό θα περιπλέξει τα πράγματα ιδιαίτερα στις μικρές χώρες, θα αυξήσει το διοικητικό άχθος, θα χρειαστούν, ε, θα χρειαστούν ε, περισσότερες προσπάθειες για τον συντονισμό. Κατόπιν έχουμε το θέμα των ε, οικονομικών φορέων, των ε, επαγγελματιών. Θα πρέπει αυτοί να λαμβάνουν μέτρα για την εξάλληψη ε, επιβλαβών οργανισμών. Ε. Αυτό όμως μπορεί να αποδυναμώσει το καθεστώς περιγείας των φυτών, διότι η καραντίνα δεν είναι οικονομικό θέμα, δεν είναι θέμα του οικονομικού τομέα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κρατικές διοικήσεις. Το βασικό επιχείρημα για να λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς σε αυτά τα μέτρα είναι ότι οι ε, κρατικοί φορείς ε, δεν έχουν ε, επαρκείς πόρους. Οι οικονομικοί φορείς, οι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν όμως επίσης προβλήματα. Λαμβάνεται υπόψη ότι σε μικρές χώρες το 95% των οικονομικών φορέων είναι μικροί είναι μικρές ε, επιχειρήσεις, αλλά ότι η παραγωγή τους ε, είναι πολύ μεγάλη και σε μικρές χώρες ε, έχουμε περισσότερο εισαγόμενα προϊόντα και εμείς ως αρμόδια αρχή διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση της υγείας των φυτών στη χώρα μας έχει επιδεινωθεί και γι' αυτό υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Οι επαγγελματίες λοιπόν, οι εκμεταλλεύσεις αυτές ε, δεν ε, θα ε, υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους και ανησυχούμε σχετικά με την κατάσταση αυτή. Όσον αφορά τις εισαγωγές, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις απαιτήσει τις προϋποθέσεις για τις εισαγωγές. Τι γίνεται εδώ λοιπόν, τι καθεστώς δημιουργείται, θα γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι εισαγωγών. Οι εμπειρογνώμονές μας όμως πιστεύουν ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι κάπως γραφειοκρατικό θέμα, αλλά αν ε, κοιτάξουμε τον κανονισμό αυτόν, καταλήξαμε ότι ε, θα επιβληθεί τεράστιο διοικητικό άχθος ε, για την εκπόνηση εκθέσεων. Φοβούμαστε ότι οι περισσότερε προσπάθειε θα κατευληθούν για την υποβολή εκθέσεων παρά για τον έλεγχο τη υγεία ε, των φυτών, διότι ε, η, η, μπορώ να βάλω άλλου να γράψουν τι εκθέσει, αλλά δεν θα είναι εμπειρογνώμονε στον τομέα του. Ε, ε, θα θέλαμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτό το κομμάτι του κανονισμού. Ε, σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση αυτή λοιπόν ε, ήταν μια σύνοψη των θέσεων των εμπειρογνωμόνων μας. Ε, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε εργασία σας. Ε, Ευχαριστούμε Κριστίν Κιάγκο. Δίνουμε τώρα το λόγο στον Πασκάλ Παρισό, διευθυντή του τμήματος της Διεθνής Επιστημονικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Καλημέρα κύριοι βουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω την προοπτική αυτή για τα φυτά της Ευρώπης ως εκπρόσωπο της ΑΝΣΕΣ, του Εθνικού Οργανισμού της ε, Υγείας των Φυτών, της, ε, του Περιβάλλοντος και της Εργασίας. Μεγάλο οργανισμό σήμερα στη Γαλλία που καλύπτει το σύνολο των καταναλωτών, όλων των κινδύνους όπως εκτίθεται ένας ε, καταναλωτής λόγω διατροφής στο εργασιακό περιβάλλον και στο περιβάλλον. Καλύπτει λοιπόν και τα προϊόντα των φυτογενομικών προϊόντων. Καλύπτει και την υγεία των ζώων και την υγεία των φυτών. που ελέγχονται στα δικά μας εργαστήρια. Δύο λόγια λοιπόν για να σας πω το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται αυτή η προοπτική μας για την υγεία των φυτών στο πλαίσιο αυτής της κανονιστικής μεταρρύθμισης ε, ο οργανισμός μας, η ANSES, ε, συμμετοχή έχει στις ερευνητικές εργασίες ουσιαστικά για να τροφοδοτεί με στοιχεία την ανάλυση κινδύνων ε, για το σύνολο των τομέων που ανέφερα ο οργανισμός παρέξει στάσει για την προστασία υγείας στους διαχειριστές των κινδύνων στα αρμόδια υπουργεία για τη γεωργία, την υγεία, την εργασία, ενημερώνει και συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση. Ο οργανισμός μας ε, δραστηριοποιείται επίση ε, στα ε, κτηνοτροφικά φάρμακα και στο δικό μου τμήμα έχουμε 11 εργαστήρια που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης σημείο πολύ σημαντικό που θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα για την υγεία των φυτών. Να σας πω μερικά νούμερα. Έχουμε 800 εξωτερικούς ε, ειδικού που συμμετέχουν σε πάνελ εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των κινδύνων. Και η μισή ε, από τους ε, απεσταλμένους μας, τους εντεταλμένους μας εργαζόνται σε εργαστήρια για την υγεία των φυτών και των ζώων. Επιμένω σε αυτό διότι η παρουσίαση της Κομισιόν φέτος ε, αυτού του ρυθμιστικού πακέτου για την υγεία των φυτών των ζώων με το σχετικό κανονισμό για τους ελέγχους επιτρέπει να αναδειχθούν οι συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ της διαχείρισης και της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία των φυτών και των ζώων και της υγείας ε, γενικότερα των ανθρώπων διότι πολλά θέματα υγείας ε, το προερχόνται από θέματα υγείας των φυτών ή των ε, ζώων ή από θέματα υγείας που αφορούν τα προϊόντα για την ε, κτηνοτροφία ή τη γεωργία. Κάτι σημαντικό είναι ότι ο οργανισμός ε, εντάσσεται σε ανοίξει ευρωπαϊκό περιβάλλον, συνεργάζεται στενά με την ΕΦΣΑ και άλλους οργανισμούς των κρατομελών. Εργάζεται λοιπόν στους διάφορους τομείς ε, για τους οποίους έχει αρμοδιότητα με τους διάφορους ε, σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Για την υγεία στην εργασία, την υγεία του περιβάλλοντος, την υγεία των φυτών και την υγεία των ζώων. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε πολλές σχέσεις με ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς ε, αναφοράς. Μιλάμε για αναφορά που βασίζεται σε ανάλυση. Δεν αφορά ακόμα σήμερα την υγεία των φυτών. Θα επανέλθω σε αυτό. Αναφορά επίσης ε, για την επιτήρηση, διότι βλέπουμε ότι η Ευρώπη και σίγουρα η Γαλλία εργάζεται σκληρά σήμερα. Όλοι έχουν, σημεία, έχουν ανάγκη σημεία αναφοράς, για σημεία αναφορά σήμερα. Η για το ε, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και δυσκολία διαχείριση των κινδύνων. Όταν μιλάμε για υγεία των φυτών, μιλάμε για υγεία των δασών μας, υγεία των κήπων μας, υγεία των καλοπιστικών μας φυτών, μιλάμε για υγεία των δημητριακών. Μιλάμε δηλαδή για πολλά διαφορετικά θέματα, μιλάμε για... έντομα, για βακτήρια, για ιούς, ε, ορισμένα διαδίδονται από έντομα. Μιλάμε για πολλά παθογόνα. Ο κατάλογος τους πρέπει να ενημερώνεται πολύ τακτικά, ανάλογα με τα εμφανιζόμενα παθογόνα. Τα παθογόνα αυτά πρέπει να ανιχνεύονται σε κορμούς δέντρων, σε φύλλα ή σε ρίζες ή σε σπόρους. Η υγεία των φυτών λοιπόν είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Σήμερα πολλοί είναι οι κανονισμοί εκτός από τον κανονισμό και την υγεία των φυτών για τον οποίο συζητάω σήμερα και οι οποίοι είναι σημαντικοί. Υπάρχει και ο κανονισμό για του ελέγχου που επεκτείνεται στο τομέα των φυτών. Έχουμε λοιπόν ένα νέο ρυθμιστικό πακέτο σε ένα νέο πλαίσιο. Μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι έντομα που καταφτάνουν με εξωτικά φρούτα εγκαθίστανται στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Σημαίνει επίσης ότι ορισμένα μανιτάρια λόγω της κλιματικής αλλαγής αναπτύσσονται πιο εύκολα στα δημητριακά ε, και ενέχουν κινδύνους ε, για την ανθρωπινή υγεία. Μη κοιτάς τέτοιοι. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν επηρεάζει σημαντικά την εγκατάσταση και ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών, ε, καραντίνας που μέχρι σήμερα δεν επιζούσαν όταν εισάγονταν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η διατροφική ασφάλεια πολύ σημαντικό για 9 δισεκατομμύρια κατοίκους περισσότερο από ποτέ πρέπει να διατηρούμε, να προστατεύουμε την ασφάλεια και την υγεία των φυτών ώστε να αποφεύγονται οι σπατάλες ε, λόγω επευλαβών οργανισμών. Και τέλος ε, έχουμε τις νέες χρήσεις στον τομέα των φυτών. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από φαντασία το περιβάλλον μας, ακόμη και το αστικό περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς τύπους καλλιεργιών. Τώρα έχουμε και τείχους ε, και σκεπές ε, φυτών, όλα είναι δυνατά. Κάθε φορά που έχουμε λοιπόν μια νέα πρακτική έχουμε νέα φυτά που μπορεί να εισαχθούν στην επικράτειά μας. Όταν μιλάμε για καλοπιστικά φυτά, μίλαμε και για, και για πιθανά ζυζάνια στη Γεωργία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μπορούμε να τα διαχειριστούμε αρμονικά με ικανή παραγωγή, ικανοποιητική παραγωγή και προστασία της υγείας. Εγώ αποφάσισα να πω 70 χρόνια καθυστέρηση που πρέπει να καλύψουμε Εάν συγκρίνουμε με την κτηνιατρική και τις γνώσεις των παθογόνων και τις επιδημιολογίες τους στον κόσμο των ζώων, όπου ο αριθμός των παθογόνων είναι πολύ χαμηλότερος, η υγεία των φυτών έχει καθυστερήσει πολύ, παρότι μιλάμε για αλυσίδες υψηλής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας Στο σημερινό περιβάλλον γνωρίζουμε πολύ καλά τις αρνητικές συνέπειες ορισμένων μορίων ε, προϊόντων φυτοϊγειονομικής που απαιτούν για την υγεία των γεωργών και των συμπολιτών μας να μειώσουμε τη χρήση ε, φυτοφαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να διαγνώσουμε πολύ προσεκτικά τι παθογόνα υπάρχουν και από ποιο επίπεδο μόλυνσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέτρα αντιμετώπισης για τις καλλιεργίες. Ε, μετά τον πόλεμο η χημεία μας επέτρεψε να αυξήσουμε τις αποδόσεις μας σημαντικά χωρίς τις ανησυχίες που έχουμε σήμερα διότι τότε δεν γνωρίζαμε ακόμα τη χημεία τόσο καλά όσο τη γνωρίζουμε σήμερα. Οι άνθρωποι πέθαναν νωρίτερα, συνεπώς δεν είχαμε όλες τις παθολογίες που εμφανίζονται λόγω των χημικών προϊόντων που οφείλονται σε αυτό φάρμακα, αλλά και μόνο. Μιλάμε και για τα πρόσθετα πλαστικά και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η γνώση που έχουμε στην τοξικολογία και στη χημεία θέτουν σε αμφισβήτηση τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την προστασία μας και την υγεία των φυτών μας ε, τρέφοντας τον πλανήτη αλλά προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Τέλος, νομίζω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη, στα περισσότερα προσέχουμε ιδιαίτερα το δημόσιο χρέος και τους οικονομικούς περιορισμούς που βαρύνουν τα κράτη-μέλη. Καλό είναι λοιπόν να, εργαζόμαστε αποδοτικά και να περιορίζουμε την εισαγωγή παθογόνων. Πώς θα γίνει αυτός ο περιορισμός ε, με διατάξει περιορισμού των εισαγωγών και του εμπορίου, περιορισμό και των δραστηριοτήτων των ιδιωτών, διότι όταν ε, μπαίνουν νέα φυτά, αν είναι φυτά στο μπαλκόνι μας δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά αν τα φυτά αυτά μπουν σε ένα κήπο κοντά σε καλλιέργειες, τα πράγματα γίνονται πιο σημαντικά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η αξιοπιστία των διαγνώσεων. Είναι απαραίτητο τα εργαστήρια αναλύσεων να κατέχουν τις επαρκείς ικανότητες ε, με σωστή ρύθμιση. Αυτό υπάρχει για, την... για τον Υπάρχει μια αλυσίδα εργαστήριων σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να επιτευχθούν οι στόχοι του αναθεωρημένου κανονισμού ώστε να είναι πιο αποδοτική η δημόσια Να υπάρχει δηλαδή μια λίστα που θα ενημερώνεται τακτικά ώστε τα κράτη-μέλη να μην σπαταλούν χρόνο σε παθογόνα που δεν υπάρχει πλέον λόγος να παρακολουθούνται να έχουν ευελιξία, να χρησιμοποιούν είτε ανταλλαγή μέσων μεταξύ των κρατών μελών ε, και ανταλλαγή μεθόδων ανάλυσης ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις μας το να διασφαλίζεται η συνοχή των δράσεων και αυτό πρέπει να αποτελεί στόχο του κανονισμού και το επίπεδο δράση με μέτρα προσαρμοσμένα στους κινδύνους. Και συχνά οι διαχείριστες των κινδύνων έχουν την επιλογή του μέτρου διότι είναι τόσο πολλοί αριθμα τα παθογόνα που είναι δύσκολο να δοθεί ένα μέτρο που να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αντιδραστικότητα τώρα και αξιοπιστία, τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω, ανάπτυξη της επιτήρησης που σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου στον τομέα της υγείας των φυτών ε, και που απαιτεί μέσω της μοριακής βιολογίας να παρακολουθούμε ε, τις αιστείες που, από προέρχονται και πώς κυκλοφορούν. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης αποτελούν κομμάτι του σχεδίου κανονισμού. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια σχέδια μόνο για τα παθογόνια. Τα σχέδια των κρατομελών πρέπει να καλύπτουν τις καλλιέργειες, τις καλλιέργειες καλοπιστικών φυτών και τα δάση. Διότι τα μέτρα θα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τομέα. Διάλογος με τους διαφορούς φορείς είναι πολύ σημαντικό. Για να καλύπτουμε όλους το μίσο από τη διάγνωση μέχρι την επιτήρηση. με την εικόνα που έχω εγώ για την υγεία των φυτών και την υγεία των ζώων, πιστεύω ότι αυτό το ρυθμιστικό πακέτο και ειδικά αυτό ο κανονισμό για την υγεία των φυτών αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να καλύψουμε το κενό και να αναπτύξουμε την υγεία των φυτών ε, σε επίπεδο αντίστοιχο με τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και του περιορισμού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Πασκάλ Παρισό. Το λόγο έχει ο κ. Κλάου Ράκ. πρώτος τον κύριο Σιλβέστρης ε, ήθελα να υπενθυμίσω να καλέσω τους εμπειρογνώμονες μας να περιορίζουν στα 10 λεπτά το χρονομιλία τους ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει συζήτηση και απάντηση στις ε, ερωτήσεις ε, που θα θέσουν οι συνάδελφοι. Σας καλώ λοιπόν, παρακαλώ να περιοριστείτε σε 10 λεπτά. ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μισή ώρα διαθέσιμη για τη συζήτηση. Κλάους Ραφ. Κλάους Ραφ, μέλος του... Μέλος ε, της ε, Κιβωτού του ΝΟΕ, ο κύριος ε, Κλάους Ραφ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλβέστης. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου παρέχετε να σας παρουσιάσω την προοπτική για την βιοπικιλότητα είναι μουσιακή αυτή η ας το πω χαρακτηριστική μορφή ή είναι κάτι που θα διασφαλίσει τις επιστικές ανάγκες της ανθρωπότητας στο μέλλον. Γεύσεις, χρώματα, απόλαυση με... Ε, την οργάνωση από την οποία προέρχομαι που είναι μια ένωση εδώ και πάνω από 20 χρόνια με αυξανόμενο αριθμό ε, μελών. Έχουμε ένα κήπο οργανικής καλλιέργειας, 6.500 ε, είναι εκείνοι οι οποίοι ε, είναι οι δυνατότητες πρόσβασης στην τράπεζα σπόρων. Έχουμε ένα δίκτυο σπόρων, έχουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκπαίδευση και κατάρτιση. Τι είναι η βιοπικιλότητα. Είναι γενετική βιοπικιλότητα παρέχοντας δυναμικές διαδικασίες ορίμανσης στο χρόνο. Δυναμικά, δυναμική διαμόρφωση σχήματος, γεύσεων, ε, ποικιλότητα στην, ε, στις δυνατότητες μαγειρικής και ε, μαγειρεύματος. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Τα χρειαζόμαστε διότι η γενετική βιοπικιλότητα είναι η βάση της ίδιας της ύπαρξής μας για εμάς και τη ζωή μας είμαστε οι ε, θεματοφύλακες αυτού του σημαντικού θέματος που διασφαλίζει τη ζωή μας. Και έχουμε εδώ και τα δίκτυα των ίδιων των γεωργών και καλλιεργητών. Τι γίνεται λοιπόν με την ε, ποικιλότητα. Αυτό που βλέπετε αριστερά καταδεικνύει μόνο μία ποικιλία που αποκαλείται ε, καΐμπι πιπεριά και είναι, ας το πω έτσι, ε, έχει σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο για ε, να υπάρξει μια ε, σταθεροποίηση σε σχέση με το προτινόμενο νομικό πλαίσιο απαιτείται η δυναμικότητα, δηλαδή να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες περιβαλλοντικές. <clears throat> Τι είναι αυτή η ποικιλότητα, μια και διαρκώς μετεξελίσσεται και μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των φυτών μπορεί να υλοποιήσει τον προτινόμενο ορισμό ποικιλότητα όπως έχει προταθεί. Το να είναι κάτι σταθερό και ε, ομοιόμορφο δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για αυτά τα φυτά. Ποια καλύτερη ρύθμιση νομοθετικά μπορούμε να αναμένουμε υπάρχει δραματική διεύρυνση του φάσματος από 250 είδη που θα μπορούσαν σε 300.000 είδη να επεκταθεί ε, το νομικό πλαίσιο στην οικουμένη. Ένα τεράστιο βάθος και εύρος νομοθετικών διατάξεων σε κάθε φάση που θα απαιτείται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο. Πρέπει να δούμε σε σχέση με την αύξηση αυτή όσα προβλήματα συνδέονται στοχεύει και θα έπρεπε να στοχεύει και να ρυθμίζει μόνο την εμπορική εκμετάλλευση των ε, ε, σπόρων των φυτών που είναι ένα, ένας άλλος ε, χαρακτηρισμός της επαγγελματικής δραστηριότητας ε, καθώς επίσης και άτυπα συστήματα ε, σπόρων και όλες τις άλλες ε, δραστηριότητες που δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα που θα έπρεπε να αποκλείονται. Στο σημερινό σύστημα μόνο οι εμπορικές εταιρείες καταχωρούνται. Υπάρχει όμως ανάγκη μαζικής καταχώρησης. Όλοι οι γεωργοί που θα έχουν σχέση με σπόρους, οι έμποροι, λιανικής, οι καλλιεργητές, οι βελτιωτές, οι κυπουροί θα έχουν υποχρεώσεις να καταχωρούνται και να να Το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρχει μόνο μία δεδομένη προδιαγραφή στην οποία θα πρέπει νομοθετικά να ανταποκρίνονται όλοι οι άλλοι. Και έτσι βιομηχανικά φυτά ε, όσον αφορά την ανταπόκριση θα μπορούν να ε, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ο γενετικός πλούτος ε, μέσα σε μία ποικιλία δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Και ο αριθμός των ποικιλιών όσον αφορά την αύξηση ετήσια θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει πολύ μικρός ε, βαθμός ε, διαγενετικής ποικιλότητα, ε, χαμηλός βαθμός όσο αφορά τα σπουδαιότερα είδη και δεν είναι ευχολόγιο, δεν είναι κατάλογος βάση με το, του οποίου θα μπορεί κανείς να αγοράζει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε τέτοια ποικιλία. Τι βλέπουμε λοιπόν, απώλεια βιοποικιλότητας. απώλεια ποικιλότητας κατά τα τελευταία 100 χρόνια. 75% απολέστηκε η ποικιλότητα και έχουμε κιόλας ε, και πάνω από 100 χρόνια ε, έντονη καλλιέργεια. Τυχαία είναι όλα αυτά. Θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι διαθροτικές αλλαγές στη γεωργία. Αλλά επίσης ε, η εισαγωγή περιοριστικών διατάξεων για την εμπορία αυτών των φυτών και σπόρων που επιβάλλεται στον αριθμό των εμπλεκόμενων στην αγορά που περιορίζει πολύ σημαντικά τα πράγματα. Ένα ισοδίκιο πλαίσιο δραστηριοτήτων μπορεί να προσεγγιστεί με διαφορετικό τρόπο. Το σύστημα της καταχώρησης ποικιλότητας και αδειοδότησης παρεμποδίζει την πρόσβαση στην αγορά για νέους ε, ενδιαφερόμενους ε, που θέλουν να ε, εμπλακούν σε αυτή την αγορά και βλέπουμε ποια προβλήματα υπάρχουν ήδη σε αυτή την αγορά. Να φανταστούμε ένα συγκρίσιμο σχέδιο με τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις σε άλλες δραστηριότητες, για τα εστιατόρια για παράδειγμα. Τι θα γινόταν εκεί. Θα έπρεπε μια συνταγή κάποιου μάγειρα να καταχωρείται σε μια αρμόδια αρχή προτού μπορεί να μαγειρεύεται ένα πιάτο. Θα έπρεπε να διαχωρίζεται από άλλες συνταγές. Θα πρέπει να είναι ενιαία η συνταγή με συγκεκριμένες ποσότητες και φυσικά θα χρειάζεται αδειοδότηση, πιστοποίηση. Θα πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια αρχή για την οποιαδήποτε προσαρμογή αλλαγή της ε, μαγειρικής συνταγής. Θα συγκρίνονται όλα αυτά τα στοιχεία σε σχέση με την αρχική συνταγή και θα έχουμε και ελέγχους για την πιστοποίηση όσον αφορά το μαγείρεμα. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να φανταστεί πώς θα επλήττονται οι μάγειροι και οι μαγειρικοί ε, από τέτοιου είδους ρυθμίσεις ένα σύστημα <clears throat> ποικιλία, ε, προστασίας ποικιλιών υπάρχει ήδη. Δεν χρειάζεται ένα τέτοιο νέο σχέδιο περιοριστικό το οποίο θα δημιουργούσε de facto ένα νέο πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τώρα, αναπαραγωγικό φυτικό υλικό. Εδώ διακυβεύεται αυτό. Όχι, δεν υπάρχει καμιά σχέση με την αλυσίδα τη διατροφική. Διότι το αναπαραγωγικό υλικό δεν το βάζουμε στο στόμα μας, το φυτεύουμε στο έδαφος. Και όταν έχουμε τέτοιου είδους καλλιέργειες, εκατομμύρια τέτοιες ε, ε, διεργασίες ε, ολοκληρώνονται και πολλές από αυτές δεν μπορεί κανείς να τις έχει όλες υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε το καλύτερο νομοθετικό έργο και η ρύθμιση να διαμορφωθεί για τις ανάγκες μας. Ζητάμε να υπάρχουν θεμητοί και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού που θα βασίζονται σε ισοδίκαιο πλαίσιο δραστηριότητα από πλευρά των καλλιεργητών και των ε, βελτιωτών. Να υπάρχουν κίνητρα για τους μικρογεωργούς, να μειωθεί η επιβάρυνση και τα προσκόμματα, να μειωθούν και όχι να αυξηθούν. Να διασφαλίσουμε διαφάνεια, για ένα καθεστώ διαφάνεια για εκείνου που θέλουν να γνωρίσουν ποιε μέθοδοι και ποια πλαίσια είναι στη διάθεσή του. Επίσης, οι διαφορετικοί τρόποι, τα διαφορετικά υποδείγματα, πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με αυτή τη γεωργική προσπάθεια για την αηφορία. Όλο και περισσότερο επικεντρωνόμαστε στην ΚΑΠΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική και άλλες πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου <clears throat> θα πρέπει με τέτοιου είδους άξονες να, να, καθορίσουμε τη δράση μας. Η βιοπικιλότητα είναι μια αρχή που ισχύει στην φύση. Δεν είναι ένας προστατευόμενος τομέας δραστηριοτήτων είναι η παγκόσμια οικουμενική αρχή, αρχή που ισχύει στη φύση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να αποφύγουμε την υπονόμευση της βιοπικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς υποχρεώσεις που επομίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ανταγωνισμός διατάξεων λοιπόν και ρυθμίσεων, ο οποίος θα είναι αναγκαίο επακόλουθο αυτής της νομικής ρύθμισης, θα έχει υποχρεωτικές καταχωρήσεις και αδειοδοτήσεις. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Θα πρέπει να είναι θελοντικό το πλαίσιο αδειοδότησης πιστοποίησης και μετά η ίδια η αγορά θα κάνει τις καλύτερες επιλογές. Υπάρχουν καλύτερες επιλογές για τους χρήστες, ε, όπως αυθεντική πραγματική ελευθερία να επιλέγει κανείς από πολυάριθμους, ε, ε, από μεγαλύτερη προσφορά προϊόντων, παραγωγών και καλλιεργητών. Η διαθεσιμότητα των πιο σπάνιων και οικονομικά μη σημαντικών καλλιεργειών θα αυξηθεί και η διαφάνεια για τις μη παραδοσιακές ε, μεθόδους παραγωγής ε, θα μπορέσει και αυτή να ε, κατοχυρωθεί. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερες επιλογές για τους καταναλωτές και για τα ασπάνια και παραδοσιακά φυτά. Θα είναι ασφαλή αυτά, γιατί για όλα αυτά τα φυτά και όσα απορρέουν από αυτά, το επίσημο με συγχωρείτε, η επίσημη αρχή για τους ελέγχους θα εφαρμόζει τις ε, αναγκαίες διατάξεις. Αν είχαμε μια νομοθεσία σαν αυτή που προτείνεται τώρα, σήμερα, την είχαμε πριν από 11.000 χρόνια, δεν θα είχαμε τη γεωργία και δεν θα είχαμε μετεξελιχθεί και αναπτυχθεί εδώ που φτάσαμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Κλάους Ραπφ και δίνω τώρα το λόγο στον καθηγητή Ρομπερτο Πάπα, διευθύντη του Συμβουλίου Έρευνας και Πειραματισμών Γεωργίας της Φόντζα. Παρακαλώ. Uh, Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Διευθυντής ε, του κέντρου που εργάζεται για το σκληρό σύτο. Θα ήθελα να εστιάσω την παρουσίασή μου στις ε, ποικιλίε αυτές γιατί νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Όταν μιλάμε για ετερογενείς ε, ποικιλίε, μιλάμε κατά βάση για δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση αφορά τη χρήση των γεών, δηλαδή τοπικές ποικιλίε που παράγονται από τους αγρότες ε, χωρίς βελτίωση των φυτών. Μετά κάτι παρόμοιο που, στο οποίο συμμετέχουν ε, αγρότες ε, μπορεί να παραχθεί μια διασταύρωση μεταξύ διαφόρων ποικιλιών και να δημιουργηθούν διάφορα υβριδικά είδη από διασταύρωση των διαφόρων ποικιλιών. Αυτός είναι ένας τρόπος διατήρησης της ποικιλομορφίας και ανάπτυξης νέων ποικιλίων ε, στην κλασική βελτιωσή των φυτών, αλλά η εστίωση της προσέγγισης ε, της ε, βελτιώσης των φυτών και της διατήρησης των γεών είναι η έννοια της δυναμικής διατήρησης που μπορεί να διατηρήσει εξελικτικές δυνατότητες και να εστιαστεί στην προσαρμογή των υλικών, στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα σύνθετης διασταύρωσης σκληρού σύτου που δημιουργείται με τη σύνθεση διαφόρων υβριδικών ειδών, με διάφορες διασταυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα πρόγραμμα με αγρότες βιολογικών καλλιεργειών για την παραγωγή νέων ποικιλιών για βιολογικές καλλιέργειες. Αλλά αυτές οι ποικιλίες... Ε, δημιουργούνται με αυτού του είδους τις ε, δραστηριότητες. Η διαχείριση αυτών των ειδών είναι πολύπλοκη. Αυτό το παράδειγμα το βλέπει το συνάδελφο από το Μομπελιέ ε, και μετά το άλλο σημείο είναι ότι ε, τι εννοούμε όταν λέμε προσαρμογή. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε στην Αιθιοπία για το κρυθάρι. Όπως βλέπετε Το εύρος είναι από 1798 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 2855. Έχουμε τεράστιες ψωμετρικές διαφορές και όπως βλέπετε γενετική σύνθεση. Εδώ βλέπετε τους γενότυπους, τους, ε, συγγνώμη, τα τις γενετικές ομάδες με τα διάφορα χρώματα. Η γενετική σύνθεση αυτών των υλικών όπως βλέπετε αλλάζει ε, εντυπωσιακά ανάμεσα στα διάφορα υψόμετρα. Αυτό είναι σαφής ένδειξη της προσαρμογής. Γι' αυτό τον λόγο η, προσαρμογή, η προσέγγιση αυτή της εξελικτικής ε, βελτίωσης των φυτών προσαρμόζει τα φυτά στο περιβάλλον. Αυτό, ειδικέ δραστηριότητε δεν έχουμε μόνο στην Ιθοπία αλλά και στην Ιταλία όπως για την ντομάτα ή για, στην Ευρώπη για το καλαμπόκι. αποτελεί την πηγή γενετικών ε, ποικιλομορφιών και δυνατότητων προσαρμογής. Αυτές οι φυλές, ε, αυτά τα land races, αυτές οι γενετικές ποικιλίε ε, αποκτούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά το επίπεδο ποικιλομορφίας που υπάρχει εντός αυτών των πληθυσμών σε επίπεδο γεωργών, σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο χωρών είναι τεράστιο. Η ποικιλία λοιπόν, αυτά τα υλικά είναι δομημένα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με πληθυσμούς, με ε, εκτάσεις, με περιφέρειες, με χώρες. Αυτές οι δομές γίνονται με διάφορα εργαλεία. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα το δραστηριοτήτων στη Σαρδινία για το Κρυθάρι και εδώ βλέπετε ισχυρή δομή όπως στην Αιθιοπία παράλληλη με τις Αιθιοπίες, παρόμοια με τις Αιθιοπίες όπου φαίνονται ενδείξεις προσαρμογής αλλά κοιτάξτε εδώ το ποσό γενετικής παραλλαγής μεταξύ πληθυσμών είναι μόνο 14% αυτό σημαίνει ότι το 86% της ποικιλομορφίας σε όλη τη Σαρδινία βρίσκεται εντός ε, μιας ίδιας έκτασης αν θέλουμε να καταμετρήσουμε αυτή την ποικιλομορφία μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τις ποικιλίε. Η ποικιλομορφία που έχουμε στη Σαρδενία μπορεί να συγκριθεί με την ποικιλομορφία δύο στοιχειών ή έξι στοιχείων, ποικιλιών δύο στοιχείων ή έξι στοιχείων. Αυτή είναι βασική έννοια για να αναπτύξουμε ένα σύστημα για να διακρίνουμε τα είδη, τις ποικιλίε μεταξύ τους ε, είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Δεν λέω ότι είναι αδύνατον, αλλά είναι εξαιρετικά περίπλοκο και σε κάθε περίπτωση πολύ ακριβό. Ένα άλλο θέμα όμως είναι κρίσιμη σημασία για τις ποικιλίε ε, των φυτών. Οι γενετικές αυτές οι ποικιλίε ε, δεν διατίθενται από μεγάλες εταιρείες ή άλλους, αλλά ήδη οι καλλιεργητές είναι εκείνοι που τις παράγουν χρόνο με χρόνο μέσα στο χρονικό διάστημα. Και αυτό δίνει το δυναμικό για προσαρμογές. Αν λάβουμε υπόψη το να καλλιεργεί κάποιος κάτι σε ένα σημείο μόνο, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτά τα, αυτές τις ποικιλίε σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο ίδιος ο, ο καλλιεργητής ή και μέσα από άλλες δραστηριότητες θα είναι σε θέση να καλλιεργεί σε συγκεκριμένα χωράφια και εκτάσεις αυτό το υλικό. Αλλά σε κάποιο σημείο αρχίζει η εμπορία αυτών των ε, ποικιλιών. Αρχίζει η εμπορία, η διάθεση στην εμπορία αυτών των γενετικών ποικιλιών. Και λέει κάποιος, ωραία, να το κάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε τώρα να καλλιεργούμε αυτή την ποικιλία και να την διαθέτουμε στο εμπόριο. Έτσι χάνουμε μεγάλο βαθμό βιοποικιλότητας. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά Ποιε επιπτώσει θα έχει ένα τέτοιου είδου σύστημα, ποιε επιπτώσει θα υπάρξουν με τέτοιε αλλαγέ στην νομοθεσία. Οι πτυχέ λοιπόν αυτέ τη αγορά μπορεί να είναι σημαντικέ για να βοηθήσουμε κάποια ανταλλαγή στοιχείων και γνώσεων μεταξύ γεωργών στο τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσε όμως ε, να είναι μια πολύ σημαντική περιπλοκή αν έχουμε την ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών από πλευρά τους και εγκαταλειφθούν οι παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Σαν συμπέρασμα, συμπερασματικά, τρία σημεία θέλω να τονίσω. Το πρώτο, η δυναμική ε, διατήρηση συντήρηση είναι πολύ σημαντική ε, ως στοιχείο και μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ε, φυτοπλασμάτων και σπόρων και αν διασφαλίσουμε το δυναμικό για προσαρμογές θα έχουμε την δυνατότητα να αυξηθούν αυτά τα φυτά και ε, θα έχουμε την δυνατότητα να οριμάζουν και θα αν δεν προσέξουμε την ε, διαφοροποίησή τους μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όταν θα έχουμε μόνο μια ενιαία εμπορία. Πρέπει αυτά να διασφαλιστούν ως βιοπικιλότητα. Να χρησιμοποιηθούν δυνατότητες ε, κατοχύρωσης της ποικιλότητα. Να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική αυτή η διασφάλιση ε, ποικιλότητα ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε αυτά τα είδη και να έχουμε την δυνατότητα να αποκομίσουμε τα πιο θετικά ωφέλη. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για αυτό το, το, θέμα της αγοράς θα πρέπει να το προσεγγίσουμε υπό διαφορετικά πρίσματα και να συνδέσουμε αυτή τη δυνατότητα ανταλλαγής υλικών που υπάρχει ενδυνάμει ως στοιχείο στην ομοθεσία και να δούμε πώς μπορεί να αποτελέσει επίκεντρο της δράσης μας. Είναι δυνατόν να ανταλλάσσεται αυτό το υλικό αλλά θα ήταν χρήσιμο αν υπάρχει και κάποια βοήθεια ή συμβουλευτική δράση στους γεωργούς ώστε να είμαστε ενεργά να εμπλακούμε στην συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητας ε, και να υπάρχει ε, το, να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, ποικιλο, της διαφοροποίησης των ε, ποικιλοτήτων Φαίνεται ότι δεν είναι ανέφικτο να υπάρξει ένα σύστημα καταχώρησης ε, και πιστοποίησης. Έδωσα ένα ολόκληρο πλέγμα αναφορών, αλλά υπάρχει και άλλη μία πτυχή που θα ήθελα να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την ε, αγρο ε, την πρόσθετη αγροτική αξία από αυτές τις δραστηριότητες. Βλέποντας ότι υπάρχουν αυτές οι αλλαγές τώρα σε σχέση με την πρόταση αυτή από πλευράς του εισήγητου, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, να σας θέσω ένα ερώτημα. Ίσως ε, υπάρχει κάτι το οποίο εγώ δεν αναγνώρισα που θα έπρεπε να γίνει. Γιατί την αγρονομική αξία των ποικιλωτήτων, την αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο και δεν βασιζόμαστε στο γεγονός ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό ομοιόμορφο πλαίσιο ε, με την αναγκαία διαφοροποίηση από πλευράς των καλλιεργητών χωρίς να επιβαρύνονται με περιορισμούς και διατάξεις. Έχουν αναπτυχθεί οι γεωργοί από την εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σε θέση πιθανότατα να επιλέξουν και μεταξύ διαφορετικών ε, ποικιλιών. Αυτές οι πληροφορίες και η ενημέρωση για την αγρονομική αξία των προϊόντων, των φυτών, των σπόρων είναι κάτι το οποίο πρέπει να στηριχθεί να, ώστε να αποφύγουμε, ας το πω τις μη, ε, τις μη βέλτιστες καλλιέργειες. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι αυτά είχα να σας πω και ολοκλήρωσα. Δίνω τώρα το λόγο στον Τόρ Κρέφελντ, πρόεδρο της WPC Κόπερ Τζέκα. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ, Τόρ Κρέφελντ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για το πώς βλέπουν το θέμα αυτό οι γεωργοί και τι χρειαζόμαστε στο μέλλον. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πρότασή της την προσπάθεια αναθεώρησης της νομοθεσίας για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Είχαμε ίσως την καλύτερη ε, νομοθεσία στον κόσμο το 1953 και μετά και έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σιλβέστρης για την έκθεση του που αποτελεί, μήνυμα προς τη, που αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μια εικόνα του τι σκέφτονται οι γεωργοί. οι προκλήσει προς τους γεωργούς. Πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι το 2050 θα πρέπει να ταΐσουμε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Επίσης ε, χρειαζόμαστε υψηλή ποιότητα, τρόφιμα, ζωοτροφέ και σπόρους ε, σε ανταγωνιστικέ τιμέ, διότι το 95% των γεωργών αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, πρέπει να ανταγωνιστούν δηλαδή τις παγκόσμιες τιμές. Και Η πολιτική μας ζητάει να παράγουμε και ενέργεια από τα φυτά, ενώ ταυτόχρονα μας ζητάτε ε, να ε, έχουμε λιγότερο ε, αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δηλαδή λιγότερα λιπάσματα και λιγότερα φυτοφάρμακα ανά κιλό τροφών, ζωοτροφών ή σπόρων. Έτσι λοιπόν είναι ίσως καλύτερο να μειωθεί ε, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ε, στη συμβατική γεωργία αντί ε, να μετατρέψουμε το 2% της γεωργίας σε βιολογική. Και επίσης αν κοιτάξετε ε, την ε, κατάσταση στην Ευρώπη, όλοι οι γεωργοί χρειάζονται ε, υψηλότερο εισόδημα για να κινητοποιηθεί η οικονομία στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Αλλά εάν κοιτάξουμε την απόδοση τα τελευταία δέκα χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό ε, σημαίνει και απώλεια ε, του, ε, της ανταγωνιστικότητας στον οικονομικό τομέα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Θα, πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τους ε, σπόρους. Ε, βλέπετε αύξηση της απόδοσης ε, από τη δεκαετία του 1960, αλλά την τελευταία δεκαετία δεν έχουμε αυξήσει πολύ την παραγωγή. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για κάτι τέτοιο. Μία από τις χώρες αυτές αντιπροσωπεύεται με, πολύ... με μαύρη γραμμή η Δανία. Έχει μειωθεί η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων κατά 30%. Ε, επίσης ε, οι ε, εκπομπές φόσφορου έχουν μειωθεί κατά 30% και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%. Επίσης έχουν μειώσει κατά 50% τη χρήση φυτοφαρμάκων. Υπάρχουν τεχνολογικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Ένας από τους λόγους όμως είναι ότι ε, χρησιμοποιεί 90% νέων ποικιλιών κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό σύστημα καταχώρησης. Οι γεωργοί γνωρίζουν πώς μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τους σπόρους που θέλουν. Κάθε ε, περιφέρεια στην Ευρώπη μπορείτε να δείτε ε, τι ε, ποικιλίε παράγει, ε, τι γίνεται με τους συμβατικούς γεωργούς, τους βιολογικούς γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους χειροτρόφους. Μπορεί λοιπόν να εισάγει ο γεωργός την καλύτερη ποικιλία για την δική του περιφέρεια. Επίσης μπορεί να δει σε τι βαθμό μπορεί να μειώσει τον, τη χρήση μη κοιτοκτόνων. Ε, μπορεί επίσης ε, να δει Μπορεί επίσης ε, να δει την ανθεκτικότητα στους μήκητες, στην ξηρασία κλπ. Ε, ίσως λοιπόν στις δοκιμές VCU καλό είναι να συμπεριλάβουμε και άλλα στοιχεία ώστε οι γεωργοί να γνωρίζουν τι αγοράζουν διότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αυξηθεί το εισόδημα των γεωργών. Όταν δηλαδή ο γεωργός γνωρίζει ότι θα έχει καλή απόδοση από τους σπόρους που θα φυτέψει. Ε, το, η δοκιμή VCU λοιπόν, ε, αξίας καλλιέργειας χρήσης, ε, αποτελεί ε, πολύ καλό ε, εργαλείο για τους γεωργούς. Ο γεωργός γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει με αυτό το τεστ. Προτού εισαχθεί αυτό το σύστημα γινόταν πάντα συζήτηση ανάμεσα στους βελτιωτές των σπόρων και τους ε, γεωργούς. Ε, ε, δεν ήξερε ποια είναι η ποιότητα των σπόρων. Το 1953 όμως, κατόπιν αιτήματος των γεωργών, εισήχθη η νομοθεσία και έκτοτε η ποιότητα των σπόρων βελτιώνεται κάθε χρόνο. Και αυτή τη στιγμή που εκπονείται τη νέα νομοθεσία λέμε ότι θέλουμε η υψηλότερη ποιότητα σπόρων. Θέλουμε οι βελτιωτές ε, να ε, βελτιώσουν περαιτέρω ε, τις ποικιλίε, διότι η Ευρώπη χάνει έδαφος στον ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό διότι έχουμε πολλούς γεωργούς στην Ευρώπη πολλών διαφορετικών ειδών. Έχουμε τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, έχουμε τις συμβατικές και έχουμε τις βιολογικές. Δεν μπορούμε ε, στην δοκιμή VCU να ελέγξουμε τις βιολογικές ποικιλίε για βιολογικούς στόχους. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους βιολογικούς σπόρους και τους άλλους, διότι ε, πρέπει να... Διότι στη συμβατική γεωργία έχουμε τα χημικά προϊόντα που μας βοηθούν. Πρέπει λοιπόν να ε, εξεταστούν οι σπόροι αυτοί από την οπτική της βιολογικής γεωργίας. Και όταν εξετάζονται οι σπόροι για τους στόχους αυτούς, ε, μπορεί ο Γιώργος ε, να είναι βέβαιος ότι αυτή η ποικιλία θα είναι η κατάλληλη για αυτόν. Τέτοια πράγματα ζητάμε λοιπόν. Επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν συστήματα καταχώρησης στην Ευρώπη που λειτουργούν ε, καλά. Ανέφερα το δανέζικο σύστημα, υπάρχουν όμως και άλλα στη Γερμανία, στην Αγγλία και αλλού. Πρέπει να διαδώσουμε το ότι όλοι οι γεωργοί, ιδιαίτερα στις νέες, στα νέα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες ε, σχετικά με το τι είναι καλή ποικιλία για τον ίδιο τον γεωργό διότι οι γεωργοί στην Κόπα Κοσέγκα ε, ανησυχούν ότι ανοίγουμε ε, την πύλη για μια μεγάλη αγορά ότι θα εισαχθούν στην αγορά πάρα πολλοί σπόροι οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Πολλοί γεωργοί σε κάποιες ε, χώρες ε, χάνουν, ε, εξαπατώνται διότι τους πολλούν σπόρους των οποίων τις ιδιότητες δεν γνωρίζουν. Ο μόνος λοιπόν που χάνει εδώ πέρα είναι ο μικρός γεωργός και έχουμε 2 3 εκατομμύρια τέτοιων στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να τους λάβουμε και αυτούς υπόψη μας. Κατόπιν φτάμε στο ετερογενές υλικό που δεν είναι ούτε ποικιλία ούτε μείγμα ποικιλιών διότι ε, όπως έχει αυτή τη στιγμή η πρόταση της Κομισιόν ξέρουμε ότι θα έχουμε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα ε, αποκαλέσουν το υλικό τους ετερογενές υλικό και θα μπορέσουν έτσι να εξαπατήσουν τους γεωργούς. Αυτό όμως ε, δεν είναι καλό για τους γεωργούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιο υλικό. Σας ε, ζητούμε λοιπόν να φροντίσετε να βρείτε μία λύση ώστε αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιο υλικό να έχουν την απαραίτητη αγορά αλλά να μην μπορεί ο καθένας να υποφεληθεί από την αγορά αυτή. Ε, οι εξειδικευμένες αγορές. Ε, μια παλιά ποικιλία δεν είναι εξειδικευμένη, εξειδικευμένος τομέας της αγοράς. Έχουμε κάποιες ε, μη επαγγελματικές ενώσεις που θέλουν διατήρηση των ε, διαφόρων ποικιλιών. Ε, εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για την αγορά που απευθύνεται στους επαγγελματίες. Οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί εξειδικευμένη αγορά, εξειδικευμένο προϊόν, ε, ακόμα και κάποιες από τις παραδοσιακές ποικιλίε, εάν είναι υψηλής ποιότητας, ε, ε, μπορεί να θεωρηθεί εξειδικευμένο προϊόν, αλλά δεν θα είναι εξειδικευμένο εάν υπάρχουν πολλοί παράγοντες στη συγκεκριμένη αγορά. Και επίσης από την πλευρά των γεωργών έχουμε πολλά μέλη που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όταν ε, μιλάμε για τέλη. Μπορεί να μιλάνε για 50 ευρώ, έχουμε όμως 150 ε, ευρώ. Έχουμε 2 ή 3 εκατομμύρια γεωργών στην Ευρώπη, για τους οποίους 150 ευρώ το χρόνο είναι ε, σημαντικό ποσοστό του εισοδήματό του. Όταν λοιπόν μιλάμε ε, για τέλη, φροντίστε και οι μικροί γεωργοί να μπορούν να επιβιώσουν και να μπορούν να αγοράσουν σπόρους υψηλής ποιότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε τώρα τον λόγο στον Γκάρλι Καρονέσεν από το European Seed Association για 10 λεπτά και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τι ερωτήσει έχουμε χρόνο μέχρι τις 6 και μισή διότι μετά οι δερμηνείς πρέπει να αναχωρήσουν. Έχουμε λοιπόν περιορισμένο χρόνο, 10 λεπτά λοιπόν ομιλία τώρα και μετά μας μένουν 35 λεπτά πριν για τη συζήτηση. Έτσι πολύ. Λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ Γκαρλή Φωνέσεν. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά να παρίσταμε εδώ απόψε ανάμεσά σα συνειδητοποιώ ότι πιέζει ο χρόνος και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πέντε διαφάνειες έχω όλες και όλες που θα σας δείξω. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τη συζήτηση και έτσι θα βοηθήσω να είμαι και σύντομος στην παρέμβασή μου, συντομότερος. Ο τίτλος είναι απλός. Δυναμικό για ανάπτυξη. Potential for growth. Αυτό βλέπουμε από προτάσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δυναμικό για να υπάρξουν ακόμα και βελτιώσεις του ήδη ισχυρού δυναμικού του αναπαραγωγικού τομέα και της παραγωγής φυτών στην Ευρώπη και να παρέχουμε τα βέλτιστα προϊόντα και ήδη ώστε να μπορέσουν οι γεωργοί μας να καλλιεργήσουν εκείνα τα οποροκυπευτικά και προϊόντα που χρειάζονται και πρέπει. Δεν θα επιστέθω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί έχετε και στοιχεία και σημειώσεις από τη γραμματεία που σας έχουν παρασχεθεί για τη δομή του ευρωπαϊκού τομέα σπόρων και κάποια από αυτά τα στοιχεία αναφέρονται και στις διαφάνειες. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι κάποιους μύθους καταργούν και ακυρώνουν. Δεν υπάρχει κάτι σαν λίγες μεγάλες εταιρείες που να δεσπόζουν παγκόσμια η εικόνα είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη. Εξαρτάται από τι καλλιέργειε, από τη χώρα, από τα είδη, από τι ποικιλίε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διακύμανση και ποικιλία. Ναι, υπάρχει επικέντρωση και συγκέντρωση όπω σε οποιονδήποτε άλλο οικονομικό τομέα στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν ο τομέα των καλλιεργειών και των σπόρων να εξαιρείται. Είναι ένα υψηλή τεχνολογία τομέα. Εργαζόμαστε με τεχνολογία και επιστήμη εχμή. Και όλα αυτά κοστίζουν ε, μεγάλα κονδύλια, πολλά χρήματα. Είναι λοιπόν φυσική αυτή η κατάσταση. Όμως, όπως πληροφορηθήκατε από τη γραμματεία, πολύ λιγότερο υπάρχει δεσπόζων ρόλος στην Ευρώπη από κάποιες λίγες μεγάλες εταιρείες από ό,τι σε σχέση με άλλες χώρες και η ε, και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει αποτελεσματικότητα αυτού του νομοθετικού πλαίσιου που συζητάμε σήμερα, που παρέχει και διασφαλίζει ένα ισοδίκαιο πλαίσιο δραστηριότητας. Αντικειμενικές δυνατότητες για τους γεωργούς να συγκρίνουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Και έτσι ταυτόχρονα παρέχεται η ευκαιρία για μικρές εταιρείες να υποφεληθούν από το γεγονός ότι τα προϊόντα τους ε, θα είναι, μπορούν να είναι καλύτερα από εκείνα των μεγάλων μεγαλύτερων ανταγωνιστικών εταιριών. Αυτοί είναι οι πυλώνες ε, της σημερινής, ε, ας το πω έτσι, πρότασης αναπαραγωγής στην Ευρώπη των, της Seed Marketing Legislation, της ε, διάθεσης στην αγορά των σπόρων, η ταυτότητα των προϊόντων, τι εμπεριέχεται σε ένα σακουλάκι από πλευρά σπόρων, η ποιότητα των σπόρων, το δυναμικό και οι επιδόσεις αυτής της ποικιλία σπόρων στο ίδιο το χωράφι, τι μπορεί να παράξει μια τέτοια ποικιλία σπόρων και προφανώς και οι απαιτήσει για την υγεία. Η διασφάλιση δηλαδή ότι οι σπόροι που φυτεύουν οι γεωργοί θα είναι ελεύθερες από οποιασδήποτε επιμολύνσεις. Αυτή είναι η πυλώνες λοιπόν. Αυτοί οι πυλώνες ε, ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς οδήγησαν τον ευρωπαϊκό τομέα σπόρων να γίνει ένας από τους πρωτοπόρους, τους προπομπούς παγκόσμια, στην παγκόσμια σκηνή. Και το είδαμε αυτό. Όμως υπάρχουν και προσεγγίσεις που συμμερίζονται όλοι οι χρήστες του αναπαραγωγικού υλικού των σπόρων. Άσχετα αν είναι κανείς γεωργός μεγάλης κλίμακας ή αν βρίσκεται σε μια αγορά νης εξειδικευμένης διαχείρισης και δραστηριότητας ή αν δραστηριοποιείται σε άλλες ποικιλίε. Αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε να διασφαλιστεί είναι το υλικό, να γνωρίζουμε τι είναι το υλικό που χρησιμοποιούμε, να γνωρίζουμε ότι η ποιότητα αυτού του υλικού είναι αυτό που αναμένουμε και προσδοκούμε, ότι έχει τις επιδόσεις στο χωράφι που προσδοκούμε και ότι δεν θα είμαστε θύματα των ε, ασθενειών. Αυτοί λοιπόν οι επιτυχείς πυλώνες διασφαλίστηκαν και διατηρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Και εμείς από πλευρά του τομέα μας τονίζουμε και απευθύνουμε έκκληση σε εσά να διατηρήσετε, να διατηρηθούν αυτοί οι πυλώνες. Ήταν τα ειχέγγυα, ο θεματοφύλακα τη επιτυχία που σημείωσε αυτό ο τομέα στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν και κάποιε ανησυχίε που έχουμε σε σχέση με αυτή την πρόταση. Υπάρχουν ένα αριθμό εξαιρέσεων. Υπάρχουν αρκετέ εξαιρεσει, ε, απαλλαγέ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι εμπορία που προβλέπονται. Και δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ποια θα είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών σε συνδυασμό μεταξύ του. Συζητήσατε σήμερα το πρωί για παράδειγμα το θέμα του ποιος θα καλύπτεται, ποιος είναι ένας επαγγελματίας στην επαγγελματική του αυτή δράση, σε αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη των εμπόρων σπόρων ότι πρόκειται για την διάθεση στην εμπορία αυτού του αναπαραγωγικού υλικού. Δεν πρόκειται για ανταλλαγή απλώς μεταξύ κυπουρών ή μικρογεωργών κάποιων σπόρων είναι διάθεση στην εμπορία με επαγγελματικό τρόπο από επαγγελματίες εταιρείε λοιπόν που εισπράττουν, αποκομίζουν έσοδα και κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό είναι ο πυρήνα η καρδιά αυτή τη νομοθετική πρόταση. Και συμφωνούμε με αυτήν και αυτή είναι η καρδια αυτη τη νομοθετικη προταση και συμφωνουμε με αυτη και αυτη ειναι η ουσια η ουσία αυτής της πρότασης. Ίσως όμως ε, δεν είναι απόλυτα σαφής ε, αυτή η δυνατότητα ορισμού και ίσως πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, διευκρινήσεις. Το δεύτερο είναι οι πολλές εξαιρέσεις και απαλλαγές για τις δυνατότητες νίσια, για το ετε, ετερογενή υλικά, για τις διαφορετικές ποικιλίε. Έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι έγινε μια προσπάθεια να παρασχεθούν ευκαιρίες για πολύ συγκεκριμένες αγορές και τις ανάγκες τους αυτή η απόπειρα όμως, αυτή η πρωτοβουλία περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και καθιστά ακόμα δυσχερέστερη την κατανόησή τους και πρέπει και το συνειδητοποιούμε αυτό να υπάρξουν βελτιώσεις σε αυτό το πλαίσιο. Χρειαζόμαστε και ένα μέσο, ένα εργαλείο σαν αυτό που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περιγραφή των στοιχείων και στόχων. Ένα εργαλείο και μέσο που ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πάνω από ένα από τα στοιχεία αυτών των αγορών. Υπάρχει μια ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε εχέγγυα για την ενημέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών, να έχουν οι καταναλωτές κάποια στοιχεία, όμως να μειωθεί, να απαμβληνθεί η διοικητική επιβάρυνση για εκείνους που δεν θέλουν να ακολουθήσουν την κλασική ε, νομοθετική διαδικασία και τις κλασικές διαργασίες ε, διασφάλισης ε, και καταχώρησης αυτών των ποικιλίων. Αναφέρθηκε πολλές φορές το κατόφλι 10 απασχολούμενων για εταιρείε που βρίσκονται εντός του πλαισίου και θα καλυπτόντουσαν από αυτήν την νομοθεσία. Εμείς διαφωνούμε με αυτό το πλαίσιο. Εγώ θα έλεγα αν ήμουν υπεύθυνο για μια εταιρεία που θα είχε τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ και κάποιους λίγους απασχολούμενους δεν θα σκεφτόμουν ότι είμαι απλά ένας ερασιτέχνης. Ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν. Αυτός ο τζίρο εκατομμυρίων δείχνει, καταδεικνύει ότι είμαι επαγγελματίας και ότι αποκομίζω κέρδη από αυτή τη ε, δραστηριότητά μου. Δίκαιο και σωστό αυτό, αλλά δίκαιο και σωστό αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτέ τι δραστηριότητε να υλοποιούν ελάχιστε προποθέσει. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με έναν αποκλεισμό. Θα συμφωνούσαμε με κάποιε προσαρμογέ όσον αφορά τις διατάξει και του κανονισμού. Τελευταία παρατήρηση για την ιχνηλασιμότητα, την ανείχνευση και την ε, διασφάλιση διαφάνεια στο συνολικό σύστημα να αποκατασταθεί έτσι η εμπιστοσύνη. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτέ τι αγορέ έναντι των πελατών του υποχρεούνται να διασφαλίζουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαφάνειας. Τι σημαίνει αυτό. Πράγματι σημαίνει απλά νομοθετικά πλαίσια. Να είναι κάποιος επαγγελματίας, ο οποίος πολύ επαγγελματικά αυτού του είδους τα προϊόντα ως υλικό στους πελάτες του. Δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι υπερβολικό ως απέτηση, ούτε χρειάζεται να πει κανείς ότι αυτό είναι ιδιαίτερο πρόσκομα ή γραφειοκρατικό εμπόδιο. Αλλά τούτων λεχθέντων Παράλληλα με όλα αυτά βαίνει και η ανάγκη της σωστής ετικετοποίησης και επισήμανσης ε, από πλευράς ε, της ε, συσκευασίας. Να γνωρίζει ο πελάτης που αγοράζει αυτά τα προϊόντα, αυτούς τους πόρους, να έχει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να του διατίθενται, άσχετα αν ασχολούμεθα με την επαγγελματική αγορά, με επαγγελματίες ή αν ασχολούμεθα με κάποια εξειδικευμένη δραστηριότητα που αφορά συγκεκριμένες διαχειριστικές πράξεις έναντι άλλων εναντί τρίτων. Όλα πρόκειται, αφορούν την εμπιστοσύνη λοιπόν στο τέλος τέλος. Δεν θα βλέπουν κάποιους πόρους και θα επαρκεί αυτό για να ξέρουν οι άνθρωποι ποιο προϊόν θα ε, φυτρώσει από αυτούς τους πόρους. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα να γνωρίζει ο γεωργός αν αυτό το υλικό παραχθεί και φυτευτεί μέσα σε αυτό το σύστημα με αυτούς τους όρους θα έχω την προσδοκία να παράξει και να φυτρώσει με τον τρόπο που αναμένεται και προσδοκούμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν το πλαίσιο εμπιστοσύνη από πλευρά συστήματος. Κατανοούμε ότι αυτό απαιτεί και μια ελαστικότητα, μια ευελιξία. Η ελαστικότητα ή η ευελιξία δεν πρέπει όμως να υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ανέφερα αυτή την πρόταση, αυτή τη διατύπωση στο τέλος. Η μελλοντική νομοθεσία πρέπει να προαγάγει την καινοτομία, να προάξει επίσης ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, να διασφαλίσει πλαίσια ασφάλειας για τους γεωργούς, αλλά να δημιουργήσει και ένα πλαίσιο ισοδίκαιας δραστηριότητας για τους, υπογραμμίζω εδώ, επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτό τον τομέα. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, τότε για να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που αναφέρθηκαν απόψε, τότε πράγματι η αναθεώρηση θα έχει επιτύχει τους στόχους της. Η μεταρρύθμιση αυτή νομοθετικά θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα, θα μειώσει τις δαπάνες και τα έξοδα για τους γεωργούς και καλλιεργητές αλλά και για τους πελάτες τους. Και συνολικά <clears throat> θα είναι ένα καλύτερο σύστημα από εκείνο που χρησιμοποιούσαμε και είχαμε στο ε, παρελθόν, πέρα από το ότι θα υπάρχουν και ε, ε, οι ανάγκες εξοικείωσης. Αν τα καταφέρουμε θα είναι μεγάλη επιτυχία που θα στέψει αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ και για τις προτάσεις σας ε, και τα κίνητρα που δώσατε στο τέλος. Έχουμε τρεις συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν, Ντόρφ, Ρόσλινγκ και Άνιου. Συνάδελφους Ρόσλινγκ και Άνιο. Να τους δώσω το λόγο αμέσως για τις παρεμβάσεις τους και τυχόν ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων. Στο τέλος ε, θα δώσουμε το λόγο για λίγα λεπτά στον συγγνώμη, στο τέλος θα έχουν όλοι οι προγραμμονές 3 με 4 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα ακούσουμε. Παρακαλώ, συνάδελφος κ. Ντόρφμαν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα για τις τελευταίες παρεμβάσεις και στους τελευταίους που παρενέβησαν όσον αφορά τους σπόρους και το αναπαραγωγικό υλικό να πω ότι όλα αυτά τα θεώρησα πολύ ενδιαφέροντα σίγουρα θεωρώ ότι οι τέσσερις εισηγήσει ήταν άκρος ενδιαφέρουσες και κατέδειξαν κάτι το ότι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο διαφορετικά πράγματα έχουμε εδώ ενώπιόν μας που δεν πρέπει να συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Το ένα, το πρώτο είναι, αν επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, η κλασικής μορφής γεωργία, άσχετα αν είναι παραδοσιακή ή άλλη μορφής γεωργία όπου εκατομμύρια γεωργών, γυναίκες και άνδρες σε εκμεταλλεύσεις γεωργικές πανευρωπαϊκά παράγουν τρόφιμα για τις αγορές. Πολύ καλά. Όποιοι το κάνουν αυτό και δραστηριοποιούνται έτσι, όποιοι σπέρνουν σπόρους ή φυτεύουν, για παράδειγμα, πατάτες ή αμπέλια ε, ή έχουν άλλες καλλιέργειες και δασοκομική δραστηριότητα. Πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις που θα μπορούν να τηρηθούν για αυτούς. Και μετά υπάρχει μια άλλη αγορά, μια άλλη αγορά που την αποκαλούμε δραστηριότητα νης ίσως, δραστηριότητα συγκεκριμένων ε, διαχειριστικών δράσεων ή δραστηριοτήτων, όπου με μεγάλη ικανοποίηση καλλιεργητές, ε, κάποιες ποικιλίε που έχουν, τις καλλιεργούν και παράγουν προϊόντα εντός εισαγωγικών πιο ε, παραδοσιακά σε μικρές αγορές ε, ή μικρότερες αγορές που έχουν κάθε λόγο ύπαρξης ε, και δικαιολογούνται να υφίστανται. Ο κανονισμός για τον οποίο συζητούμε εδώ δεν είναι ο ενδεδειγμένος να έχουμε ιδεολειπτικά έναν πόλεμο ε, ιδεολογικό, τι είναι καλύτερο, τι είναι χειρότερο από τα δύο. Και για τα δύο είδη γεωργίας πρέπει να βρεθούν οι σωστότερες λύσεις. Εντάξει, και θα έλεγα ότι οι επαΐοντες, οι πραγματογνώμονες διαφοροποιήθηκαν επαρκώς επ' αυτών ώστε να, να ληφθεί αυτό το στοιχείο υπόψη. Απλά κάποιες ερωτήσεις θα είχα. Προς τον πρώτο για την εισήγηση του κυρίου ε, Ραφ. Τι μας είπε ο κύριος μα είπατε ότι στον τομέα εφαρμογής αυτού του κανονισμού εντάσσονται κάποιοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο. Αναφέρεστε προφανώς στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3, όπου αναφέρεται στο 2, για παράδειγμα, ότι στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μόνο επιχειρήσεις και εταιρείε εντάσσονται. Μα εταιρείε, οι επιχειρήσεις είναι επαγγελματικής δραστηριότητας εταιρείε. Έχετε μία άποψη πώς καλύτερα νομοθετικά θα μπορούσε να ρυθμιστεί αυτό και να διατυπωθεί. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί η διατύπωση και η ορολογία. Δεν είναι ιδανική αυτή η τοποθέτηση. Τώρα, για εσάς τον δεύτερο κύριο, μιλήσατε για τις νίσες. Πώς θα καθορίζατε το θέμα των νης αυτών των διαχειριστικών ε, ή εμπορικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, είπατε για κάποιους συνεργάτες που θα είχατε ένα τζίρο εκατομμυρίων. Πώς μπορεί ένας τέτοιος, ε, μια τέτοια δυνατότητα να καθοριστεί επακριβώς. Υπάρχει κάποιος λογικός ε, ή με κοινό νου που θα έλεγα να αποσαφηνίζει τα πράγματα με την κοινή λογική. Μια πρόταση να καθορίζει την ενίσχυση τελευταίο από πλευρά ε, του καθηγητού Πάπα στην παρέμβασή του. Είπατε, συνεχίζει η Ιταλική. Είπατε, μιλήσατε για επαρκή και απαραίτητη βιομηχανία και εγώ συμμερίζομαι τη θέση αυτή. Εσείς ε, λέτε ότι που λέει ότι στην τάδε περιφέρεια χρειάζεται αυτή η, η ποικιλία, αλλά αν υπάρχει μόνο η ε, ε, τότε σίγουρα θα λέει ο καθένας ότι η δική του ποικιλία είναι καλύτερη στον κόσμο. Ποιος ορίζει τι είναι καλύτερο. θα γίνεται ε, από κάποια δημοσιαρχή. Ποιος θα το αποφασίζει αυτό. Herbert. Ευχαριστούμε Χέρμπερτ, συνάδελφος Όσλαγγ. <clears throat> Καταρχήν μια ερώτηση προς τον κύριο Κούφουτ. Επειδή η Κόπα Κοζέκα σε μια ακρόαση ανέφερε υπάρχει λέει μια μαύρη αγορά μια παραοικονομία. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η εμβέλεια αυτής της μαύρης αγοράς, να δώσετε κάποια αριθμητικά μεγέθη. Στην Ευρώπη είναι ένα λέει, ευρύ φαινόμενο αυτό ως φαινόμενο. Ακούσαμε διάφορα τι πρέπει να ρυθμιστούν κατεπηγόντως. Πιο πριν ακούσαμε όμω από την άλλη πλευρά ότι παρόλη την μη ύπαρξη κοινών κοινοτικών κανόνων <clears throat> ε, βρισκόμαστε καθοδόν με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές. Τι θέλουμε, αναμένουμε ένα μεγαλύτερο ακόμα ποσοστό σε σχέση με την, ε, τις επιδόσεις μας. Ποιο είναι το ε, εύρος, ο στόχος, ο συγκεκριμένος στόχος που θέλουμε να ρυθμίσουμε με αυτή τη δράση. Από ό,τι ε, κατάλαβα από τον προλαλήσαντα δεν επιθυμεί καθόλου να υπάρξει αγορά νης συγκεκριμένων εξειδικευμένων διαχειριστικών δυνατοτήτων. Είπε ότι όλα πρέπει να ρυθμιστούν ενιαία. Και δεν ξέρω αν με τη ρύθμιση αυτή είσαστε ικανοποιημένος, αλλά ας το πούμε έτσι, 250 διαφορετικά πράγματα, όλα, όλες οι ποικιλίε να ενταθούν σε αυτόν τον κανονισμό. Δηλαδή βότανα, χόρτα, λουλούδια, ε, δέντρα, όλα να καταχωρούνται σε ένα ευρωπαϊκό κεντρικό μητρό ή κατάλογο. Ε, ποιος θα υποφεληθεί. Θα υπάρξει τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση μόνο. Και στα όσα αναφέρθηκαν με τους συναδέλφους, ε, ε, εμείς δεν είμαστε και εμείς υπέρ μιας τέτοιας ρύθμισης. Πρέπει να μην γίνει κεντροποιημένη προσπάθεια εναρμονισμού. Να μην συγχαίουμε την προσπάθεια εναρμονισμού με μια ε, κεντρικού χαρακτήρα, με ένα κεντρικού χαρακτήρα σχεδιασμό και υπερβολικές ρυθμίσεις και περιορισμούς αναφέρθηκε κάπως γενικόλογα ότι υπάρχουν λέει κάποιοι παραδοσιακοί τομείς αλλά δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα όπως στη είπα ή σε άλλες υπήρους. Αλλά όταν έχουμε 50,5% δεσπόζοντα ρόλο στην αγορά ε, όσον αφορά το καλαμπόκι από κάποιους λίγους πέντε παραγωγούς επιχειρήσεις, πέντε επιχειρήσεις και έχουν 70% με συγχωρείτε ποσοστό της αγοράς αυτές οι πέντε επιχειρήσεις. Και αν σκεφτούμε άλλους τομείς ε, για τα οποροκυπευτικά, πέντε επιχειρήσεις 45% των της τομάτας ε, καλύπτουν και μια επιχείρηση 20% μόνη της. Να μην κάνω λόγο για όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Η τάση είναι σαφής προς επικέντρωση και προς ένταση στην εκμετάλλευση. Και δεν υπάρχει επιλογή αν τρεις μεγάλες εταιρείες έχουν στα χέρια τους το 90% του σπανακιού, της παραγωγής σπανακιού στην Ευρώπη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν απασχολεί τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη ε, ή κάποιος αντιφάσκει. Τώρα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφείς ενδείξεις ότι έχουμε επικέντρωση, συγκέντρωση, συμπίκνωση των συμφερόντων της αγοράς από λίγες επιχειρήσεις. Σε ένα μεγαλύτερο εύρος όμως ε, ε, σπόρων που θα πρέπει να εξεταστεί ως μελλοντική προοπτική ώστε για αυτές τις αλλαγές ε, που ε, επιτυγχάνονται να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα όλων. Και δεν μπορούμε έτσι να προσαρμοστούμε, δεν προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς διότι άλλοι εξωθούνται εκτός αυτής της αγοράς. Δεν υπάρχουν δυνατότητες για αυτούς. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας καλώ να είστε εκεί πιο σύντομοι, διαφορετικά δεν θα προλαμβάνω να ακούσουμε όλες τις απαντήσεις όλων των εμπρογνωμών. Συνάδελφος κύριε Σάνιο. Πρόεδρε, Πόσο μπορώ να μιλήσω. Τέσσερα λεπτά θα ήταν το ιδανικό. Ε, νομίζω θα τα καταφέρω. Τρεις ερωτήσεις, ε, δύο πολύ συγκεκριμένες. Ε, μία προς τον ομιλητή από την Αυστρία που είπε ότι υπάρχει ε, μείωση της ε, βιοπικιλότητας κατά 74% μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε ε, χίλια διαφορετικά είδη φυτών στην Αυστρία το 1917, τώρα έχουμε μόνο 240. Αυτό λέει και με όλο το σεβασμό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Ναι, κάποια Μπορεί να έχουμε μείωση κάποιων ειδών, ε, μάλλον ε, ε, ο αριθμός φυτών σε κάποια είδη μπορεί να έχει μειωθεί, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έχουν εξαφανιστεί τελείως. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με την πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση από τη Δανία. Το ότι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την ε, την παραγωγή μειώνοντας ε, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν. Ε, τι χρησιμοποιείται η βρύδια. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι η ιστορία επιτυχίας του τομέα των σπόρων. Πιστεύετε ότι έχοντας κατά νου αυτή την ιστορία επιτυχίας είναι απαραίτητη η νέα νομοθεσία διότι θα θεωρούσε κανείς ότι αφού τα πράγματα πάνε καλά, στα αφήσουμε όσο έχουν. Επίσης, πριν κάποιους ε, μήνες ε, το κοινοβούλιο μας ε, απαγόρευσε τα νεονικοτινοειδή χωρίς σωστή επιστημονική βάση. Μπορείτε να μας πείτε ότι ωραία είμαστε άνθρωποι των σπόρων, όχι των διαφόρων υλικών επεξεργασίας των σπόρων, αλλά εάν αποσυρθεί ένα προϊόν που χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία. Στην ουσία έχουμε ε, διαφορετική ποικιλία διότι ε, μπορεί ένα τέτοιο προϊόν να αντισταθμίσει μια δυναμία στην ποικιλία. Μήπως μπορείτε σας παρακαλώ να ε, σχολιάσετε το θέμα των νεονικοτινοειδών, των ουσιών επεξεργασίας των σπόρων και του Κοινοβουλίου γενικά. Η κυρία Ρόντους για να ολοκληρώσει και μετά οι επαΐοντες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ πολύ έλεγα που μου δίνετε πολύ σύντομα το χρόνο να παρέμβω. Με πολύ, έχω σύντομες ερωτήσεις μόνο. Πιστεύω όταν κάνουμε λόγο για νης, για τέτοιες δυνατότητες, δεν θα πρέπει να μιλάμε για συνεργάτες ε, και τζίρο, αλλά για τους σπόρους και το υλικό σπόρων για σπορά. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Μπορείτε να μου πείτε ότι προς αυτή την κατεύθυνση των σπόρων θα βαίνει ο ορισμός και όχι προς κατόφλια συνεργατών και τζίρου μετά κατέστη σαφές ότι όλα αυτά πολύ δαπανηρά θα είναι και θα κοστίσουν μεγάλα κονδύλια και όσον αφορά και την έρευνα και την ανάπτυξη και τα συναφή. Στο τέλος τέλος από αυτή τη συζήτηση πρέπει να απορρέει ότι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με παλαιές ποικιλίε και ξεχωριστές ποικιλίε έχουν και εκείνη το λόγο ύπαρξή τους. Και όταν άλλοι ασχολούνται με τη μαζική παραγωγή σπόρων και εμπλέκεται εδώ η έρευνα και η ανάπτυξη και η επιστήμη και αυτό είναι θεμητό. Δεν θέλω να ασκήσω επικρίσεις αλλά και τα δύο πρέπει να μπορούν να συνυπάρξουν και να υπάρξουν. Εκείνο που με ενόχλησε κάπως είναι η τοποθέτηση της κυρίας Παριζό που είπε δεν υπάρχουν λέει έλεγχοι στην ε, φυτοϊγειονομική πτυχή της καλλιέργειας και των σπόρων. Ισχύει αυτό και αν ισχύει τι σημαίνει και τι πρέπει να κάνουμε τελικά. Διότι η υγεία των φυτών πρέπει ακριβώς να παρακολουθείτε και να την εποπτεύουμε όπως και τα άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, μια πολύ σύντομη παρατήρηση μόνο. Καταρχήν το ερώτημα του συναδέλφου για τη μαύρη αγορά και σε σχέση με τους σπόρους θα με ενδιαφέρε αυτό. Να υπάρξει διαφάνεια δεύτερο Επίσης το Κοινοβούλιο και αυτή η δημόσια ακρόαση είναι ένα μήνυμα σηματοδοτεί ότι θέλουμε, επιθυμούμε και χρειαζόμαστε διαφάνεια. Στη σελίδα 5 αυτού του σημαντικού εγγράφου που μας διατέθηκε, σημείο 1, περιορισμός ανταγωνισμού όσον αφορά τους πόρους και καταλήγει στις συμφωνίες μεταξύ εταιριών που την χαρτογράφηση την καθιστά ιδιαίτερα δυσχερές εγχείρημα και υπάρχει και αυτό εδώ το φύλλο. Ίσως Κάποια αποσαφήνιση ή διευκρίνηση χρειάζεται γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, Όπω είχα πει προηγουμένω, θα δώσω το λόγο στου έξι εμπειρογνώμονε που μίλησαν μέχρι στιγμή. Σα σας παρακαλώ μόνο να περιορίσετε τι απαντήσει σα σε τρία, το πολύ τέσσερα λεπτά ο καθένα. Κριστίν και Άγκο. Παρακαλώ. Sorry, atvaino, atvainojos. Es īsti nesaprotu jautājumus par augu veselību tieši. Zito, signomi, den katalava tis erotis getin getin fiton. Den katalava tin erotis getin getin fiton. Es saprotu. Procediamo con Pascal. A συνεχίσουμε με την Pascal Παρίζο. Έχει φύγει από την αίθουσα. Δεν είναι εδώ, πολύ ωραία. Κλάους Ραπ, παρακαλώ. Μάλιστα. Μια και οι περισσότερες ερωτήσεις διατυπώθηκαν γερμανικά, ας προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω γερμανικά σε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για κάθε ερώτηση, για τη δική σας ερώτηση κύριε Ντόρφμαν. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε φυσικά προτάσεις πώς αυτοί οι ορισμοί μπορούν να διατυπωθούν με τέτοια απόλυτη σαφήνεια ώστε να είναι εύληπτοι και σαφής όπως ζητήθηκε. Συγκεκριμένη πρόταση στο άρθρο 3 εδάφιο 6. Τα υποεδάφια α έως ε να διαγραφούν ώστε να απομένει η διάθεση στην αγορά του F, του σίγμα ταφ, του στίγματος και η εισαγωγική διατύπωση να συμπληρωθεί για χρήση για την εμπορική εκμετάλλευση, commercial exploitation. Όπως μέχρι σήμερα, στις μέχρι σήμερα οδηγίες είχαμε και προβλεπόταν. Και να συμπληρώσουμε κάτι στο άρθρο 2, να διαγραφούν οι λέξεις, δύο λέξεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ούτε στο στόχο της ε, ρύθμισής μας. Τώρα, για την ερώτηση που διατυπώθηκε από την κυρία Ρόντουστ. Απάντηση ναι, μάλιστα. Και εδώ μπορούμε να φανταστούμε την αγορά, τις αγορές νης. Αλλά να μην υπάρξει παρανόηση. Νης, θέλω σωστά και δίκαια να ερμηνεύσω τις προτάσεις της Επιτροπής. Δεν αναφέρεται στο μέγεθος αφεαυτού μιας επιχείρησης ο όρος νης, αλλά αφορά συγκεκριμένη χρήση συγκεκριμένου υλικού. Δηλαδή, σε σχέση με τον ορισμό αυτού του κανονισμού να προβλέπετε ένα όριο. Γιατί διότι οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση με απλό τρόπο να κρίνουν και να σταθμίσουν περί τίνος πρόκειται, αν υλοποιούνται κάποιοι όροι και προϋποθέσεις ή όχι. Εμείς όμως θεωρούμε μία άλλη ένδειξη για εξίσου απλή, εξίσου εύκολη στη διαχείριση και επαλήθευση, δηλαδή τον, το, την ε, έκταση επί της οποίας επιτυγχάνεται η παραγωγή, η φύτευση. Θα μπορούσαμε εδώ σε σχέση με τις διαφορετικές περιφέρειες ε, ε της Ευρώπης να έχουμε συγκεκριμένα τέτοια στοιχεία ώστε από αυτές τις ε, εκτάσεις ε, όταν έχουμε παραγωγή ε, σπόρων να μπορούν αυτές οι διατάξεις για τις νης, για αυτές τις δραστηριότητες να ισχύουν. Προς τον κύριο Άγνιου τώρα, δεν έκανα λόγο για είδη, έκανα λόγο για ποικιλίε αλλά με τον παλαιό όρο, όχι με, με τη νέα έννοια που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Φυσικά είναι δύσκολο επιστημονικά να συγκρίνει κανείς ε, τέτοιου είδους πράγματα μετά την εισαγωγή ενός ε, συστήματος με το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου κανείς δεν είχε μητρώα και καταλόγους και δεν είχαμε τέτοιες καταχωρήσεις. Όμως, σύμφωνα με τις γενετικές τράπεζες και τις ε, εγγραφές και καταχωρήσεις εθνικά σε αυτές και σύμφωνα με την έρευνα όσον αφορά τις, ε, τους καταλόγους και τις επιχειρήσεις σε, διάφορα, σε διάφορες χώρες, μπορεί να συναρθεί ως συμπέρασμα ότι περίπου κατ' εκτίμηση 70% της γενετικής ποικιλότητας που υφίστατο τότε παλαιότερα όχι σε σχέση με, ε, με, με, διάφορους, ε, ε, με διάφορες ποικιλίε, για παράδειγμα γενετικές ποικιλίε, 70% έχουν απολεστεί. Δεν είναι διαθέσιμες καν, ούτε καν σε γενετικές τράπεζες σπόρων το 70% το 25% υπάρχει και <clears throat> είναι πολύ μικρότερο βέβαια αλλά το διατηρήσαμε και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αναπαραγωγικούς στόχους και για το θέμα της υγείας των φυτών φυτοϊγειονομικά θέματα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σωστή επιλογή και προσέγγιση επέλεξε να επικεντρωθεί στα ζυζάνια εκείνα τα οποία πρέπει να τεθούν υπό καθεστώς καραντίνας και δεν ανήκουν στα όσα παρατηρούνται και υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι εισαγόμενα. Δηλαδή ε, επιζήμια για τις καλλιέργειες και τα φυτά που πρέπει να καταπολεμηθούν άμεσα που σε μεγάλο βαθμό όμως με αγρονομικά μέτρα μπορούν να αντιμετωπιστούν ώστε να θεραπευτεί η κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια είδη από αυτά που είναι ιδιαίτερα προβληματικά και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ε, με εξαίρεση φυσικά την μαζική χρήση χημικών φυτο, ε, ζυζανιοκτώνων, παρασιτοκτώνων, εντομοκτώνων κτλ που ε, δεν είναι κάτι το ευκταίο. Όμως με έλεγχο να υπάρξουν βελτιώσεις είναι η βασική μας προσέγγιση και δεν μπορώ από την δική μου πρακτική ως γεωργού να πω ότι αυτό είναι το πιο ενδεδειγμένο. Όταν παρουσιαστεί κάτι πρέπει μέσα σε λίγες ώρες, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αντιμετωπιστεί και να μην σταυρώσουμε τα χέρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρομπέρτο Πάπα. Ναι. Θα απαντήσω αλλά στα γερμανικά, κύριε Μπάρθμαν, όσον αφορά τον ντους. Υπήρξα λίγο γρήγορος. Αλλά ήθελα να πω προφανώς η αξιολόγηση της αγρονομικής αξίας, δηλαδή τα, οι δοκιμές προσαρμοστικότητας των υλικών πρέπει ούτως ή άλλως να γίνονται βάση των όσων γίνονται αυτή τη στιγμή των όσων υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν καταλαβαίνω. Μια επικοινία που δεν έχει αγρονομική απόδοση, αλλά ενδιαφέρει την αγορά, διότι έχει χαρακτηριστικά αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Επειδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια αγορά, ε, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να καταχωρηθούν με όλες τις διασφαλίσεις που παρουσιάζει το σύστημα διαπίστευσης. Κυκλοφόρησε στην αγορά και τέλος, ε, λέει ο Γεωργός, ξέρω ότι αυτή η υποκειμενικα επειδη για παραδειγμα υπαρχει μια αγορα για οποιοδηποτε λογο δεν μπορουν να καταχωρηθουν με ολε τι διασφαλισει που παρουσιαζει το συστημα διαπιστευση κυκλοφορησε στην αγορα και τελο λεει ο γεωργος ξερω οτι αυτη η ποικιλια παράγει λιγότερο αλλά την καλλιεργώ διότι την αγοράζουν οι έμποροι. Η... Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός ενδιαφέροντος προϊόντος. Η μόνη αιτία θα ήταν να σκεφτούμε ότι οι αγρότες ε, βάσει των όσων λέμε εμείς δεν θα μπορούν να επιλέξουν. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται σε όλες τις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις διάφορες ε, ποικιλίε. Ε, εντάξει, υπάρχει και θέμα κόστου, που πρέπει να υποστεί ο καθένα να προσταλώνει ήταν λίγο περίπλοκα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό θα επελύει τα προβλήματα και τη εξειδικευμένη αγορά. Γιατί μια εξειδικευμένη αγορά που αύριο δεν είναι εξειδικευμένη. Ξεκινάει ω εξειδικευμένη, αλλά μετά διευρύνεται. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα σύστημα που θα διασφαλίζει μια διαπίστευση, μια επιστοποίηση. Τώρα αυτή η πιστοποίηση για την αγρονομική αξία μπορεί να μην βασίζεται σε κίνητρα. Θα πρέπει να επινοήσουμε κάτι άλλο, ανάλογα με την περίπτωση, κάτι πιο απλό. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις ε, για τη γενετική, πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Θεωρώ ότι ήταν λίγο έντονη η δήλωσή σας. Ε, σήμερα στη γενετική υπάρχουν νέες ποικιλίε, ε, για παράδειγμα στα άγρια είδη, έχουν περισσότερες αντοχές και τα λοιπά και υπάρχει και η άλλη ότι οι τοπικές ποικιλίε υπάρχουν ακόμα με μεγάλη ποικιλομορφία. Συνεπώ πρέπει να προσέχουμε όταν αξιολογούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ρομπερτο Πάπα. Τουρκέφιντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μία ερώτηση αφορούσε τη μαύρη αγορά σπόρων. Ε, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Έχουμε παράνομες εισαγωγές και μη πιστοποιημένους σπόρους. Σπόρους που εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς κανέναν έλεγχο. Και αυτό ε, με οδηγεί στο να αναφέρω όταν μιλάμε για υγεία των φυτών τη Νέα Ζηλανδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ε, εισάγεται κανένας σπόρος ε, χωρίς ε, έλεγχο. Στην Νέα δεν επιτρέπεται ούτε ένας τουρίστας να φέρει μια χούφτα σπόρους. Ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό και σε κάποιες ε, χώρες όπου δεν έχουν έναν ε, κατάλογο καταχωρημένων ε, ποικιλιών οι γεωργοί ανταλλάσσουν σπόρους, πολλούν σπόρους ένα στον άλλον και υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που βάζουν πολλά λεφτά έτσι και ποιος χάνει αν ε, ως ε, γεωργός αγοράσω πολύ ακριβούς σπόρους και τελικά έχω πολύ κακή απόδοση. Γι' αυτό στην κόπα συζητάμε την ποιότητα των σπόρων. Ο γεωργός ε, πρέπει να έχει δικαίωμα ελεύθερη επιλογή, αλλά θα πρέπει να ξέρει τι διαλέγει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα καλό σύστημα καταχώρησης, ώστε ο γεωργός να γνωρίζει τι αγοράζει. Και όταν μιλάμε για εξειδικευμένες αγορές, τι είναι οι εξειδικευμένες αγορές ε, και στην κόπα συζητιέται πολύ αυτό. Υπάρχουν πολύ μικροί γεωργοί, βρίσκουν μια ποικιλία, υπάρχει μια μικρή τοπική αγορά, υπάρχει κάποιο εστιατόριο που θέλει να πληρώσει ε, καλά την παραγωγή του, για να αγοράσει την, την παραγωγή του. Κοινό για αυτούς είναι ότι θέλουν να κρατήσουν ε, αποκλειστικά για τον εαυτό τους σε αυτήν την μικρή αγορά και Πολύ συχνά, εάν έχουν επιτυχία, ε, κάποιος, ε, κάποια πιο μεγάλη εκμετάλλευση, πιο επαγγελματική, ε, μπαίνουν στην ίδια παραγωγή, η τιμή μειώνεται και χάνουν. Και έτσι χάνει και αυτός που ξεκίνησε την ιδέα. Όταν μιλάμε λοιπόν για προστασία των εξειδικευμένων αγορών, ε, δεν είναι πάντα καλή ιδέα να επιτρέψουμε στον, κανένα, στον καθένα να εισέλθει σε αυτή την αγορά, διότι έτσι δεν προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν από αυτό. Ακούσαμε ε, την ερώτηση αν έχουμε καλό σύστημα καταχώρησης δεν χρειαζόμαστε νομοθεσία. Όχι, χρειαζόμαστε διότι πιο σημαντικό είναι όταν αγοράζουμε μια ποικιλία να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη θα είναι η παραγωγή, η συγκομιδή, αλλά και με τις παραδοσιακές ποικιλίε να γνωρίζουμε ε, πώς είναι η ε, συγκομιδή σε σχέση με τη χρήση ε, αζωτούχων λιπασμάτων και το θέμα είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν η νομοθεσία να εξετάσει και αυτό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι για το μέλλον το οποίο να απαντά στο αίτημα των καταναλωτών ή της νομοθεσίας, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, στην παραγωγή, μπορούμε να αποδείξουμε ε, ποια είναι η παραγωγή σε σχέση με τη χρήση ε, φυτοφαρμάκων και αζωτούχων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο Γεωργός να γνωρίζει τι επιλέγει. Ευχαριστούμε. Η τελευταία ομιλία ο κύριος Γκάλικ Φωνέσεν. Βλέποντα το ρολόι, να προσπαθήσω να τηρήσω τα τέσσερα λεπτά. Ίσως για το πρώτο σημείο που δύο φορές αναφέρθηκε στην επικέντρωση και συμπίκνωση από μια παρέμβαση και τις συμφωνίες υπό αυτό το πλαίσιο. Αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Ωραία. Με την κατάσταση όσο έχει παγκόσμια και δεν είναι πλήρης η παρουσίαση, δεν είναι η πλήρης πραγματικότητα, δεν είναι πλήρης η εικόνα που αποδίδεται έτσι. Αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι ότι υπάρχουν κάποια φυτά και κυρίως, αν μπορώ να επανέλθω σε αυτό, αγορές νης, ξεχωριστές αγορές. Αν έχετε μια σχετικά μικρή αγορά δεν θα έχετε εκατοντάδες χιλιάδες εταιριών που να επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτή τη μικρή αγορά. Κανείς δεν θα θέλει να το κάνει αυτό. Και έχουμε μεγάλες αγορές δημητριακών που πάρα πολλές εταιρείες επενδύουν και έχουμε και περιφερειακά ανεπτυγμένες τέτοιες αγορές. Είναι σημαντικό να κατανοήσει λοιπόν κανείς ότι δεν έχουμε μία ενιαία ομοιόμορφη αγορά για όλους τους σπόρους. Έχουμε διάφορες αγορές σπόρων ανάλογα με τις καλλιέργειες, ανάλογα με το αν εργαζόμαστε με, το ένα ή άλλο, με τον ένα ή άλλο τρόπο ή όχι. Ναι, υπάρχουν λοιπόν πολλές συμφωνίες και άδειες. Ναι, φυσικά υπάρχουν. Είναι ένας ανταγωνιστικός τομέας και πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες συνεργάζονται όσον αφορά τον ανταγωνισμό των μεγαλύτερων, συνενώνοντας δυναμικό, ερευνητικό δυναμικό και έρευνα και δυνατότητες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ομαδοποιήσεις ή κατηγοριοποιήσεις που συνενώνουν δυνάμεις σε κατηγορίες και πλατφόρμες για να είναι πιο αποτελεσματικές και να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Αυτές οι εταιρείε δρούν και εργάζονται σε παγκόσμια κλίμακα και ε, ανταγωνίζονται παγκόσμια. Έτσι λοιπόν, ναι, υπάρχει συμπίκνωση και επικέντρωση, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί, δεν ανησυχώ εγώ για αυτή την πτυχή. Ο τομέα δεν ανησυχεί γι' αυτό. Ούτε και οι ίδιοι οι γεωργοί, οι καλλιεργητές ανησυχούν. Ίσως κάποιοι βέβαια ανησυχούν, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάνουμε λόγο για 95% των αγορών. Εντάξει, και όπως αναφέρθηκε από πολλούς ε, σήμερα έχουν είναι ικανοποιημένοι με το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα και υπάρχει ένα άλλο τμήμα όσων εμπλέκονται στην αγορά που θέλουν ένα διαφορετικό πλαίσιο. Έρχομαι στο θέμα των νης, των ξεχωριστών ε, δραστηριοτήτων ε, και δράσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ευκαιρία για αυτούς που εργάζονται με διαφορετικού είδους υλικό και γι' αυτό κάνουμε λόγο εδώ περισσότερο. Δεν κάνουμε τόσο λόγο για αγορές, αλλά για διαφορετικού είδους υλικό ή υλικά. Πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του υλικού ή των υλικών να μπορούν να το κάνουν. Και αυτό απαιτεί εξειδικευμένους ειδικού κανόνες. Συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Ρόντουστ, αν θυμάμαι καλά. Δεν θα έπρεπε για παράδειγμα να έχουμε ένα όριο σε όγκους παραγωγής, σε επιδόσεις, σε τόνους παραγωγής και μετά να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την Ευρώπη με αυτή την προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο παλαιότερα <clears throat> σε σχέση με τις παλαιότερες ποικιλίε είχαμε προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν τέλειο το καθεστώς, το αντίθετο κιόλα. Ίσως όμως είναι μια προσέγγιση που μπορεί να αναπτυχθεί και ακόμα περαιτέρω. Υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να στραφώ σε αυτό και να επανέλθω σε αυτό, σε αυτή την παρατήρηση. Κάνουμε λόγο δηλαδή εδώ για ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ή θέλουμε δύο διαφορετικές αγορές να ε, διαμορφώσουμε. Σωστό αυτό. Παρότι το δεύτερο στοιχείο της αγοράς, το νης, η νης, διαφοροποιείται πολύ από την πρώτη προσέγγιση. Δεν είμαι ακόμα βέβαιος πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Έχουμε κάποιες προτάσεις και έχουν υποβληθεί και προτάσεις. Όμως δεν είναι ανέφικτο, δεν είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε αυτού του είδους πώς να το αποκαλέσω, αμοιβαία αποδεκτό σύστημα, ενός αμοιβαία αποδεκτού συστήματος που θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αγοράς στα πλαίσια που προβλέψαμε αλλά και θα δίνει και άλλες ευκαιρίες για το μέλλον μελλοντικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βονέσαν και ευχαριστούμε όλους τους εμπειρογνώμονες που μίλησαν. Ευχαριστώ λοιπόν και τους συναδέλφους. που αντάλλαξαν απόψεις ε, με τις ερωτήσεις του έκαναν πιο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Θα μελετήσουμε αυτή την έκθεση και σήμερα πιστεύω είπαμε πολλά ωφέλιμα πράγματα. Να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 εδώ στις Βρυξέλλες. Καλό βράδυ σε όλους.